Okay, folks, can you take your... Καλημέρα σας παρακαλώ. Καθίστε στις θέσεις σας. Ξέρω ότι όπως ε, προχωράμε θα έρθουν και άλλοι συναδελφοί, αλλά κάθε λεπτό που χάνουμε τώρα είναι λεπτό χαμένο από τη συζήτηση και έχουμε ασφαλώς πολλά να πούμε. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Για δεύτερη φορά γίνεται συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας σε αυτή την ε, εβδομάδα πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ πρώτα απ' όλα να εγκριθεί η μυρίσια διάταξη, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν ανακοινώσει της Προέδρου και μπορούμε να περάσουμε χωρίς άλλη πραδιπορία στη δημόσια ακρόαση για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι είναι προφανές προφανώς ε, πολύ σημαντικό θέμα, είναι προφανή σημασία του θέματος αυτού. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο από τη συζήτηση και καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά τον Μάριο Μόντι, ο οποίος θα κάνει την εισαγωγική ομιλία για όλο αυτό το θέμα και την σημασία του όπως την θεωρεί εκείνος. Παρακαλώ λοιπόν να λάβει το λόγο ο Μάριο, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Thank you very much, Madam Chair, for... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερο ευτυχή που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σα, για δύο λόγου καταρχά. διότι ήταν για μένα η Επιτροπή σας τα δέκα χρόνια που διετέλεσα Επίτροπος ε, η πιο σημαντική επιτροπή, έχουν περάσει βέβαια αιώνες από τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει δύο πολύ σημαντικές ακροάσεις για την επικύρωση της ε, εκλογής μου ως ε, επιτρόπου είχαν να περάσω και μερικοί από εσάς ήσασταν και παρόντες τότε και και σας θυμάμαι. Επίσης, διότι η Επιτροπή σας έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, Δραματίζει και το επιτελεί το καθήκον αυτό στον υπέρτατο βαθμό βλέπω με χαρά την έγκριση του, της δέσμης για την οικονομική εποπτεία και πιστεύω ότι μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια αντίστοιχη δέσμη για την, μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση που συζητούμε και σήμερα να διαδραματίσει εξίσου σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για τα έξι σημεία. πώς βλέπω εν γέννη το πακέτο της διακυβέρνησης και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν τα ευρωομόλογα στην υπόθεση αυτή. Εν τέλει θα αναφερθώ στον ρόλο που μπορεί το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον γενικότερο αυτό, στο γενικότερο αυτό πλαίσιο να διαδραματίσει. Οι δέσμοι, λοιπόν για τη διακυβέρνηση και συμπληρώνω ότι πολύ σύντομα θα λάβετε και τρία σύντομα άρθρα μου που φαντάζομαι θα βοηθήσουν εκείνους από εσά που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συζήτηση. Το πακέτο λοιπόν για την οικονομική διακυβέρνηση είναι κατά την άποψή μου πρόοδο, ε, συνιστά πρόοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Πάντως θα ήθελα να πω εν ολίγης, ότι διαβλέπω τον κίνδυνο, παραδόξως πως, να ε, επιβαρυνθεί αρνητικά αυτό το πακέτο από μία βραχυπρόθεσμη θεώρηση ή τάση. Και θα μου πείτε πώς γίνεται, βραχυπρόθεσμο μέσα σε τέτοιο πακέτο, δεν είναι αυτό οξύμορο. Και όμως εγώ διαβλέπω ένα τέτοιο κίνδυνο, δηλαδή... Τη στιγμή που πολύ σωστά προσπαθούν να εκριζώσουν ακριβώς αυτόν τον κίνδυνο, οι πολιτικοί θύνοντες, τον κίνδυνο δηλαδή του, της βραχυπρόθεσμης θεώρησης και λήψη αποφάσεων, ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή βλέπουμε να επιβαρύνεται όλο το γίγνεσθε με αυτήν τη βραχυπρόθεσμη αντίληψη και νοοτροπία. Γιατί σας το λέω αυτό. Διότι όσοι από εμά έχουμε κάποια ηλικία και κάποια εμπειρία, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ένας αντίστοιχος κύκλος του 96-97 που ήταν άλλωστε και στις απαρχές ή μάλλον ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και πώς, πώς το ορίσαμε αυτό, το ορίσαμε ως 3,03,0 όπως λέγανε οι Γερμανοί που ήταν ο βασικός όρος για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με τον Υπουργό των οικονομικών Βάγκελ της Γερμανίας τότε και τον οποίο ακολούθησαν και άλλοι, είχε επιβληθεί αυτός ο βασικός όρος και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή ένα βασικό, απλό όμως μήνυμα, 3% επί του ΑΕΠ, ήταν ο στόχος βάση του οποίου μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ο στόχος ποιος ήταν τότε. Ο στόχος ήταν να πείσουμε μία μάλλον δύστημη γερμανική αλλά και δανέζικη κοινή γνώμη, ε, ολλανδική μάλλον κοινή γνώμη, ότι είναι απίθανον κάποιες χώρες της Νότιας Ευρώπης, κάποιοι αντάρτες που δεν θα τηρούσαν τα οικονομικά, την οικονομική πειθαρχία θα μπορούσαν να ανατρέψουν το ευρώ και έτσι θα τους επιβάλλω το ένα υψηλότερο επίπεδο πειθαρχίας Με την επιμονή αυτή στο 3,0, μετά από αυτή μάλλον την επιμονή, αποδεικνύεται ότι οι ίδιοι γεννήτωρες του Συμφώνου Σταθερότητας, Γερμανοί και Γάλλοι δηλαδή, το 2003 όχι μόνο δεν τήρησαν τις προϋποθέσεις και τους όρους που είχαν ήδη ζητήσει, πράγμα το οποίο κακό, αλλά παρεμπόδισαν τους μηχανισμούς ελέγχου και δεν τους άφησαν στη δική τους περίπτωση να λειτουργήσουν όπως έπρεπε. Και ως εκ τούτου άφησαν πεδίο δόξες λαμπρών για χώρες άλλες όπως η Ιρλανδία κτλ. Έτσι λοιπόν σε ορισμένε περιπτώσεις και αντιλαμβάνομαι η Γερμανία ιδιαίτερος ε, και άλλες υπάρχει δίψα, υπάρχει ανάγκη ουσιαστική να ε, δουν την επιβολή πειθαρχικών μέτρων ή να επανενταχθεί στην πειθαρχία την οικονομική το σύνολο αυτών των χωρών που έχουν δείξει ε, απειθαρχή και ανάρτικη συμπεριφορά όπως η Ελλάδα και άλλες. Ναι, αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να επανενταχθει στην πειθαρχια την οικονομικη το συνολο αυτων των χωρων που εχουν δειξει απειθαρχη και αναρτητη συμπεριφορα οπως η ελλαδα και αλλες ναι αυτο σημαινει βεβαια οτι πρεπει να υπαχθουν και σε μια γενικότερη αρχιτεκτονική πειθαρχία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η βούλησή τους δεν θα είναι τόσο στεγνή και μη ρεαλιστική που τελικά να καταλήξουμε σε ένα μέτρο ή σε ένα εργαλείο επιβολής πειθαρχία το οποίο τελικά δεν θα φέρει τα επιθυμούμενα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη σημασία νομίζω πρέπει να αποδώσουμε και το Κοινοβούλιο ιδιαίτερο και θέλω επί τη ευκαιρία να σημειώσω την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφω για τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου και την ποιότητά τους. Θα ήθελα λοιπόν ιδιαίτερα να δώσω έμφαση στα εξή σημεία στις προτάσεις που έχουν κατεθεί. Λιγότερη πολιτική επέμβαση, με περισσότερη μακροπρόθεσμη ε, πειθαρχία, ευρωομόλογα για να, ή ευρωπαϊκά ομόλογα για να ενισχυθεί η πειθαρχία στην αγορά και μην ξεχνάμε η πειθαρχία απαιτεί ανάπτυξη. Λιγότερη πολιτική ε, επέμβαση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως βλέπω πιστεύει άλλωστε και η Επιτροπή σας, θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο ακόμη από το προβλεπόμενο πλαίσιο και κάποιες από τις δικές σας τροπολογίες και την άποψή μου βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση, διότι, ας μην απατώμεθα, η επιβολή των μέτρων μερικές φορές παρεμποδίζεται λόγω των εθνικών παρεμβάσεων, αλλά όχι σε επίπεδο επιτροπής όπως μερικέ φορές ενδεχομένω υποδεικνύεται στο κείμενο αυτό των προτάσεων, αλλά από το Συμβούλιο. Και στην πρόταση βλέπουμε, αν δει κανεί την τελική έκθεση της Tax Force Van δίνεται η εντύπωση ότι προσπαθούν να υποβιβάσουν τον ρόλο ε, τη σημασία μάλλον το, και το ρόλο των αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή ως συλλογικό όργανο υπό τον Πρόεδρο βέβαια, αλλά ως συλλογικό όργανο. Και εγώ που ήμουν επί 10 χρόνια επίτροπος και έχω παρακολουθήσει πολύ στενά τη λειτουργία αυτού του ε, μηχανισμού, η Επιτροπή ως συλλογικό όργανο δεν ε, εξέθεσε ποτέ τον, Υπουργό των Οικονομικών, τον Επίτροπο των Οικονομικών. Αυτό το είδαμε και στην ε, περίπτωση της Γαλλίας το 2003. Ακολούθησε η Επιτροπή ως συλλογικό όργανο της ε, θέσης του Επιτρόπου των Οικονομικών Θεμάτων, των Δημοσιονομικών Θεμάτων και τελικά το, το ΕΚΟΦΗΝ ήταν αυτό το οποίο ανέτρεψε την κατάσταση. Και μάλιστα υποχρέωσε τελικά την Επιτροπή ως λογικό όργανο και μάλιστα ύστερα από πολύ έντονες διαπραγματεύσεις και διελκυστίνδες να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Γαλλίας για το λόγο αυτό. Έχουμε λοιπόν την πειθαρχία αλλά και ανάγκη για ανάπτυξη, δεύτερος όρος. Για να είναι αξιόπιστη η πειθαρχία θα πρέπει να ενταχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο όπου θα αναπτύσσεται, όπου θα υπάρχει και ανάπτυξη οικονομική, θα προάγεται η ανάπτυξη με οικονομικά μέτρα. Και εδώ βλέπω να λείπουν τα εξή στοιχεία από την πρόταση. Ενοποίηση αφενός, επενδύσεις αφετέρου. integration και innovation, τα δύο in δηλαδή για την ανάπτυξη. Integration, ενοποίηση. Στο στάδιο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι την ανάπτυξη την γεννά κατά τρόπο τεχνητό, με τεχνητή υποστήριξη του δημοσιονομικό έλλειμμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να έχει μια τέτοια προσέγγιση. Από πού λοιπόν μπορεί να προκύψει η ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο δυναμικό και απόθεμα ε, ανάπτυξης που μπορούμε να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ενοποίηση. Δηλαδή μια κοινή αγορά που θα λειτουργεί πιο καλά. Τέτοιο πράγμα όμως δεν βλέπουμε στο πακέτο αυτό για τη διακυβέρνηση να προβλέπετε. Είναι φυσιολογικό να λείπει αυτός ο χώρος από τις προτάσεις, αυτός ο τομέας. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογικό. Όταν δούμε δηλαδή ότι οι εκθέσεις της Task Force μας λένε πως με τις προτάσεις αυτές προσπαθούμε εν τέλει να ε, καλύψουμε τελικά τον οικονομικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Όχι, δεν είναι έτσι, διότι ο οικονομικός πυλώνας της ε, ΟΝΕ ποιος είναι, η μία οικονομική ένωση, δηλαδή διαρθρωτική στερεότητα της ΟΝΕ, πλήρης ενοποίηση, για την οποία δεν γίνεται λόγος καν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή επαφίεται η υπόθεση αυτή σε μια πιο ασαφή, όχι βέβαια ασήμαντη, αλλά αρκετά ενδιαφέρουσα προοπτική της Ευρώπης του 2020 που μια μέρα θα προκύψει ενιαία αγορά οικονομική κτλ. που όμως για σήμερα δεν μας δίνει λύσεις. Αυτό που θα μπορούσε να είναι για λίγο μια κάπως ελκυστική πτυχή της οικονομικής ε, πολιτικής φαίνεται να επικρατεί έναντι αυτού του άλλου κομματιού, δηλαδή της πραγματικής οικονομικής ενοποίησης, που είναι απαραίτητο στοιχείο του ε, οικονομικού αρχιτεκτονήματος της Ευρώπης. Παρακαλώ λοιπόν ξαναβρείτε τον τρόπο να επαναφέρετε την ε, ε, ιδέα αυτή της ανάπτυξης μέσα στη δουλειά. Και η άλλη σημαντική πτυχή για την ΟΝΕ είναι η διακυβέρνηση των μη νομισματικών πολιτικών. Η πολιτική δηλαδή αυτή που βλέπουμε να καλύπτεται αρκετά καλά ε, μέσα στο πακέτο για τη διακυβέρνηση. Πλην όμως, πλην όμως, το πακέτο αυτό νομίζω ότι είναι μάλλον υπερβολικά συνδεδεμένο με τις αρχικές προτάσεις του συμφώνου, με κάποιες τροπολογίες, τροποποιήσεις, διευκρινήσεις κτλ. Χάνει όμως και πάλι την σημασία, ε, ξεχνάει μάλλον και πάλι την ιδιαίτερη σημασία των οικονομικών εξελίξεων στην Ευρώπη, ότι θέλουμε αυτές δηλαδή να αποβαίνουν εις όφελος της, ε, των μελλοντικών γενεών και να μην τις καταρακώνουν. Η διάκριση εδώ δεν έχει να κάνει με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η διάκριση είναι μεταξύ τρεχουσών δαπανών, που στόχο έχουν να ικανοποιήσουν τις Σημερινέ ανάγκε και δαπανών που έχουν σε στόχο τις επενδύσεις, δηλαδή την ανάπτυξη, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές αυτές, που θα αποτελέσουν μια σημαντική, ε, ένα σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του μέλλοντος. Και εδώ νομίζω ότι θα μπορούσε να δοθεί ε, περισσότερη προσοχή και ενδεχομένως ε, με βάση κάποια στατιστικά στοιχεία να προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι οι στρεβλώσεις σε σχέση με αυτά που βλέπουμε για την Ισπανία και την Ιρλανδία είναι ε, ε, χρήσιμο να εξεταστούν. Δηλαδή, οτιδήποτε υποτίθεται ότι θα μπορούσε ως δαπάνη κρατική να θεωρηθεί ύποπτο, ύποπτη δαπάνη, τότε θα πρέπει να, ε, θα πρέπει να απαγορευθεί ενώ η αδίποτε δαπάνη επενδυτική από τον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θεωρείται καλή. Όχι, νομίζω ότι εδώ ακριβώς είναι το λάθος το οποίο κάνουμε. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε νοοτροπία στην υπόθεση αυτή. Και καλό θα ήταν να... Το είχαμε πράξει το 96 ήδη στις απαρχές αυτού του συστήματος, ήμουν από τους λίγους που το υποστήριζαν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και εν τέλει, για να αναφερθώ και στο θέμα των ευρωομολόγων, τα οποία βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, γιατί είναι ένα θέμα μεταλλασσόμενο. Ε, παρουσιάζει δηλαδή διαφορετικούς ε, και νέους κάθε φορά λόγους, τους οποίους μπορεί να είναι ελκυστική αυτή η ιδέα. Και φυσικά δεν θέλω να προδικάσω τόσο θα πούν οι λοιποί ομιλητές, η ε, πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, Ίσως τελικά να ε, μιλάμε πια για την γέννηση των ε, ομολόγων Bowles και όχι των ευρωομολόγων, αλλά ελπίζω πρόεδρε τέλος πάντων ε, να μην προβλέπω τίποτε άτοπο για το μέλλον. το γεγονός ότι προέρχεται η ιδέα αυτή από ένα βρετανικό μυαλό, από έναν εγκέφαλο βρετανικό, ίσως τελικά μειώσει ή ενισχύσει αντίστροφα την πιθανότητα εμείς ε, της υπηρετικής Ευρώπης να ακολουθήσουμε την ιδέα αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει αυτές οι συζητήσεις, τα έχουμε δει και πρόσφατα σε προτάσεις ε, για πολιτική, οικονομική και εγώ τον προηγούμενο Μάιο σε συζητήσεις με τον πρόεδρο Μπαρόσο για την οικονομική πολιτική έδωσα το στίγμα μου θεωρώντας ότι θα πρέπει να δώσουμε και περιεχόμενο και ουσία και ευρύτητα ε, στα ευρωομόλογα. Και είχα τότε ήδη αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε πως τα ευρωομόλογα θα αποτελέσουν ε, μέσον ε, δημοσιονομικής απειθαρχίας από ορισμένα κράτη. Ακολούθησε μετά ένα πιο επιστημονικά στοιχειοθετημένο έγγραφο από τον Μπρίκελ για τα μπλε ομόλογα. Μετά ακολούθησαν άλλες ε, πολυάριθμες αναλύσεις από πολλούς ε, διακεκριμένους επιστήμονες, των οποίων ορισμένοι βρίσκονται και εδώ σήμερα. Και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει ένα άρθρο στην Κοριέρε Ντελασέρα της, ε, της Δευτέρας Δεκεμβρίου, το οποίο δίνω τώρα να σας μοιραστούμε που ακολούθησε το πολύ σημαντικό πολιτικό άρθρο στους Financial Times των Γιούρκερ και Τρεμόντι. Ουσιαστικά λοιπόν είναι γνωστό πλέον πιστεύω το τι είδου πλέον εκτήματα μπορούν να προσφέρουν ε, τα ευρωομόλογα. Ευρωομόλογα εν προκειμένου δεν θα είναι δημοσιονομικά μέσα, δεν θα είναι οικονομικά εργαλεία τα οποία θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν ε, κάποιον να βγει από τη δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα είναι σημαντικά οικονομικά εργαλεία για επενδύσεις. Και αυτά που εννοώ εγώ σε ευρωομόλογα είναι σημαντικά εργαλεία για την διαχείριση του δημόσιου χρέους. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στο γιατί η υπόθεση ότι μπορεί αυτά να φέρουν δυσμενείς συνέπειες για τις ε, χρηστές οικονομικά χώρες, δεν πιστεύω ότι θα εκπληρωθεί. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε γιατί, ακόμα και για τη Γερμανία, για να είμαι σαφής, θα είναι εποφελής η έκδοση ευρωομολόγων. Θα είναι συμφέρουσα όπως θα είναι συμφέρουσα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες ε, αντιρρήσεις που έχουν ακουστεί δεν είναι εύκολο να απαντηθούν ή να διασκεδαστούν, πλην όμως μπορούν να ανατραπούν αυτά τα επιχειρήματα. Η οικονομική ανάλυση, επισημένω, αποδεικνύει πως δεν είναι δεδομένο πως η Γερμανία θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει είτε σε ονομαστικούς είτε σε πραγματικούς το κόστος της, ε, της κρατικής χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή. Και επίση, ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι το εξή, ότι αν ήμουν εγώ τουλάχιστον Γερμανό, θα θεωρούσα ιδιαίτερα θετικό το γεγονό ότι η Φερρυπίν, ο ή καγκελάριο τη Γερμανία, επεσήμανε πολύ σωστά σε μια ε, σκληρή δημόσια δήλωση ότι θα πρέπει να κληθεί και η ιδιωτική αγορά να προβεί σε ε, θυσίες. Πολύ σωστή επισήμανση που είχε και πολύ δεινές συνέπειε στην παγκόσμια, μάλλον στην ευρωπαϊκή οικονομική αγορά. Στη συνέχεια χρειάστηκε να δοθούν ε, κάποιε διαβεβαιώσεις, ναι, θα γίνει αυτό όλα μετά το 2013 κτλ. Λοιπόν, αν υπάρχει αυτή η δομή των ευρωομολόγων, εξασφαλίζει έναν φυσιολογικό μηχανισμό μέσα από τον οποίο συμμετέχει εθελοντικά, εκούσια η αγορά σε αυτή τη θυσία. Διότι αν κάποιος είναι κομιστής ε, ομολόγων της Ιρλανδίας ή της Πορτογαλίας κτλ. μπορεί να θέλει να ξεφορτωθεί αυτά τα ομόλογα, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Χρέους ε, του δημοσίου χρέους μπορεί να τα αγοράσει στην δευτερογενή αγορά και να τα κρατήσει μέχρι ότου έρθει η λήξη τους όπου στις περισσότερες περιπτώσεις θα αποζημιωθεί για ολόκληρο το ποσό το ονομαστικό ποσό των ομολόγων. Αυτό μας δείχνει γιατί στις πρώτες περιπτώσεις μπορούμε και χωρίς ε, ε, εκρηκτικές εξελίξεις να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή της αγοράς. Ταυτόχρονα διαπιστώνω, Πρόεδρο, ότι πρέπει να κλείσω την ομιλία μου. Επίσης, λοιπόν, επίσης εξασφαλίζει πειθαρχία. Δηλαδή, τι εννοώ. Μετά τη μεγάλη αυτή αναταραχή και τη συγκίνηση που προξένησε η, η, γέννηση του Euro, σαν να ήταν μανάδες, πολλές ευρωπαϊκές αγορές έπεσαν σε λίθαργο επί 10 χρόνια. Γιατί θεώρησαν ότι μπορούν όλα να λειτουργήσουν αυτόματα. Και ξαφνικά ξύπνησαν. Εάν όμως είχαμε ευρωομόλογα εξ αρχής δεν θα είχε συμβεί αυτό. Διότι με τα ευρωομόλογα αποδεικνύεται σαφώς ότι μπορεί να ασκήσει η αγορά στο ευρώ διότι υπάρχει διάκριση μεταξύ κύριου και δευτερογενούς ε, δανείου και αυτό βέβαια αντίστοιχα ε, κατανέμεται ανάλογα με το μέγεθος των των κρατών. Και εγώ αν ήμουν Γερμανός οφείλω να ομολογήσω ότι το γεγονός και μόνο πως αρχίζει ο κόσμος να, αρχίζει, να, γράφει ε, στα, στις, εφημερίδες μήπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τελικά γίνεται, μετατρέπεται σε μια κακή τράπεζα κτλ. Θα ανησυχούσα. Κανονικά η δυνατότητα απορρόφηση αυτών των κακών, ε, κακής ποιότητας ομολόγων μπορεί να έχει ε, σαν εξέλιξη κατά τρόπο ισοδύναμο με τη θεία πρόνοια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει, να μπει στην αγορά και να απορροφήσει αυτά τα κακά ομόλογα. Ναι, αλλά και νομίζω ότι ο διοικητής της Bundesbank ήταν ακριβά σαφής σε αυτό στο παρελθόν, ε, δεν είναι αυτό σύμφωνο, δεν θα ήταν κάτι τέτοιο σύμφωνο με την χρηστή διακυβέρνηση και χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρέους και θα έχει συνέπειε βέβαια και προ τη ρευστότητα του χρήματο. Ταυτόχρονα προ την ποιότητα του ενεργητικού δεν είναι καλό αυτό και έχουμε δει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανειλημμένω ζητεί διαφύλαξη τη αξία του ενεργητικού τη. Επομένω, το άριστο αυτό πλάσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ και χρόνια έχει αποδειχθεί η αξία της, θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα ξόανο μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τα ευρωομόλογα. Μήπως θα πρέπει να το αναλογιστούμε αυτό. Και για να κλείσω. Πολύ γρήγορα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδα τις εκθέσεις και πρέπει να πω ε, ότι τις είδα εντάχει μέχρι τώρα. Ε, διαπιστώνω όμω, εάν αντιλαμβάνουμε καλά τα πράγματα, ότι έχουν κοινή αξία την εξή, ότι προσπαθείτε να εισαγάγετε περισσότερη κοινοτική μέθοδο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ νομίζω ότι είναι και το κλειδί τη αξιολόγηση του κατά πόσο η δουλειά σα είναι χρήσιμη ή όχι. Και πράγματι σα εύχομαι ε, κάθε επιτυχία. Βλέπουμε επίση ορισμένε εκθέσει στη βούληση να προσδοθεί περισσότερο ρόλο και αρμοδιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ορισμένε διαδικασίε. Αναρωτιέμαι λοιπόν εγώ πέραν βέβαια του ότι είναι φυσιολογικό ένα κοινοβούλιο να διεκδικεί περισσότερε εξουσίε, από μια αντικειμενική ε, οπτική, απ' έξω. Είναι καλό κάτι τέτοιο ή κακό. Και μπορώ να σας πω τα καλά νέα, κατά την άποψή μου, γιατί εγώ προσωπικώς ήμουν πάντοτε επιφυλακτικός ως προς έναν υπερχιλίζοντα ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων σε εθνικέ δημοσιονομικέ διαδικασίε και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σιγά σιγά να συρρυκνώνεται το πεδίο δράση των Εθνικών Κοινοβουλίων σε εθνικέ οικονομικέ δημοσιονομικέ διαδικασίε. Είναι δηλαδή υποχρεωμένα εν γέννη να ε, περιορίζονται σε ένα ανώτατο επίπεδο κατά την ε, υποβολή των τροπολογιών κτλ. Τα εθνικά κοινοβούλια δηλαδή θεωρούνται ω δυνάμει παράγων δημοσιονομικής απειθαρχίας, ιδιαίτερος δε όσο πλησιάζουν οι εκλογικές διαδικασίες. Το Κοινοβούλιο λοιπόν εδώ θα μπορούσε να διαδραματίσει τέτοιο ρόλο μέσα σε αυτό το πακέτο διακυβέρνηση. Όχι. Γιατί, διότι το Κοινοβούλιο θεσμικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσμικά δεν έχει ουδεμία ανεξουσία να επιβάλλει ή να ανατρέψει την δημοσιονομική πειθαρχία σε εθνικό προπολογισμό. Σε εθνικό προπολογισμό. Ταυτόχρονα όμω, έχει και ρόλο να διαμορφώσει μια επιλογή στον κοινοτικό προπολογισμό, πράγμα όμω, το οποίο δεν συζητεί αυτό το πακέτο οικονομική διακυβέρνηση. Άρα μεγαλύτερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω προ την αξιολόγηση των δημοσιονομικών διαδικασιών μέσα στα κράτη-μέλη είναι ένας ρόλος ο οποίος δεν μπορεί να ενέχει κίνδυνο. Πρώτη διαπίστωση. Δεύτερη διαπίστωση, θεωρώ ότι θα είναι και χρήσιμο σε ένα τέτοιο ρόλο, γιατί, διότι πάλι στον τομέα αυτό θα δούμε να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο που έχουμε δει και σε άλλου τομεί, ότι δηλαδή το κοινοβούλιο μετατρέπεται στον οίκο τη διαφάνεια. Μέχρι τώρα η υλοποίηση, η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη ήταν μια διακυβερνητική συμπεριφορά και επιλογές των κρατών μελών μέσα από το Συμβούλιο ο Τομάσο Παντοσκιόπο, ο αγαπητός ε, εκλυπών, είχε μιλήσει για το καρτέλ του εθνικισμού, αναφερόμενος στο ΕΚΟΦΗΝ. Αν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσλάβει και την εξουσία να ρίχνει φως μέσα από τις διαδικασίες που θα ενταχθούν μέσα στο πλέγμα λειτουργίας του Κοινοβουλίου, να ρίχνει φως λοιπόν σε αυτά τα ε, μυστικά παιχνίδια, ε, παιχνίδια που λένε θα σε βολέψω εγώ τώρα, στήριξέ με εσύ μετά, τότε το κοινοβούλιο θα μπορέσει να αποτελέσει και θα είναι και ορατό για τον πολίτη στο ρόλο αυτό, τον φορέα της διαφάνειας στην οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, είπατε ενδιαφέροντα πράγματα για το Κοινοβούλιο και δεν χρειάζεται ε, κατά αυτόν τον τρόπο να σας υπενθυμίσουμε ότι ξεπεράσετε το χρόνο σας. Όποιος θέλει να λάβει το λόγο παρακαλώ να το δηλώσει ε, και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο. Κάποιος άλλος, Μάριο. Η πρότασή μου η οποία συζητήθηκε χθες και είναι ενδιαφέρον στο σεμινάριο που έγινε ε, για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα καταβάλλεται το, ε, ο τόκος και σχετικά με τους διάφορους μηχανισμούς διασώσεως όπως επίσης και για τα ομόλογα ε, προέβλεπε ότι όσον αφορά το ποσό το οποίο καταβάλλεται παραδείγματο χάρη από την Ιρλανδία υπάρχει και ένα επιπλέον ποσοστό ε, για τον κίνδυνο ε, της ε, αφαιρεγγιότητος αλλά θα έπρεπε να είμαστε πιο σοβαροί και να συμπεριφερθούμε σαν επενδυτικές τράπεζες δηλαδή αν στο τέλος της περίοδου έχει καταβληθεί το κόστος για τον κίνδυνο αφαιρεγγιότητος αλλά έχει αποπληρωθεί το ποσό στο τέλος περίπου το 2% το οποίο καταβάλλεται επιπλέον επί του δανείου θα πρέπει να επιστρέφεται και έτσι θα είναι ένα εξαιρετικό καρότο και έναυσμα για να μην σταματήσει κανείς τις πληρωμές του και θα είναι και πολύ καλό για την αγορά διότι η αγορά θα αντιληφθεί ότι ε, κάποια στιγμή όταν θα αποπληρωθεί το δάνειο ενδέχεται να επιστραφεί αυτό αυτό το ποσό και θα είναι ε, σημαντικό για τις ε, αναδιαρθρώσεις των δανείων ή παρεμφερείς διαδικασίες. Υπάρχει επίσης ε, και ένα δυσμενές στοιχείο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αναφερόμαστε μόνο εις τον κίνδυνο μη αποπληρωμής αλλά εάν στο τέλος δεν υπάρχει αφαιρεγγιώτης τότε πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να περιληφθεί αυτός ο όρος εάν υπάρξει αλλαγή των ε, συνθήκων. Ε, όσον αφορά τους ε, Γερμανούς δημοσίους υπαλλήλους αντιλαμβάνουμε ότι το έχουν αντιληφθεί εγκαίρως, ε, το συζήτησαν στην Δημοσιονομική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε πολλά υπουργικά γραφεία έχει γίνει μια παρεφερής διαπίστωση οπότε ίσως λέγεται όπως και εσύ είπες ότι είναι κάτι εφικτό. Ε, υποσχέθηκα σε ορισμένους συναδέλφους ότι θα διατυπώσω μία πρόταση και το πράττω τώρα. Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό σταθερότητος, να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα αυτή για να αναδιαρθρώσει το μηχανισμό και να το ενσωματώσει ίσως τα ευρωμόλογα. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ε, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι που θα συζητηθεί σε μια δεύτερη φάση αλλά είναι μια εξήγηση άπαξ και το ανέφερε ο, Μάριο και τώρα η Βίκη είναι η πρώτη στην ε, ε, συζήτηση. Ευχαριστώ σόνα. Καλό είναι ότι όλοι προσπαθούμε να έχουμε δημιουργικές ιδέες και εγώ θα ήθελα να προσθέσω μία σκέψη ότι το υψηλό επιτόκιο δεν είναι λόγω της αφαιρεγγιότητας των κρατών αλλά λόγω του ότι δεν υπάρχει ρευστότηση στην αγορά ε, είναι μία ε, σχέση μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως. Η ερώτησή μου όμως ουσιαστικά αναφερέθηκε στο θαυμάσιο επιχείρημά σας για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και για το πόσο θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον ε, ότι όλες οι δημόσιες δαπάνες δεν είναι αναγκαστικά κακές και όλες οι ιδιωτικές δαπάνες αναγκαστικά καλές. Πρέπει λοιπόν να τραβήξουμε μια γραμμή ε, για ένα δημόσιο πρόγραμμα στη χώρα μας ε, σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητος για να αναζωογονηθεί η χώρα είναι κάτι καλό και να εξετάσουμε επίσης και την ουσιαστική επένδυση που κάνουμε στην εκπαίδευση. Μακροπρόθεσμα ποια είναι η περίοδος αποπληρωμής ε, διότι ξέρω ότι αυτό συζητήθηκε πριν τα Χριστούγεννα ή ε, θα ήθελα να ξέρω αν το ξανασκεφθήκατε και τι πιστεύετε ε, ότι ε, διότι για μένα κάθε επένδυση είναι μια επένδυση στο μέλλον και όχι μόνο στην εκπαίδευση και θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Θα ήθελα λοιπόν να έχω τις ιδέες σας από πλευράς αριθμών και στοιχείων. Είναι ίσως ε, μια εξαιρετική ιδέα να συγκεντρώσουμε διάφορες ερωτήσεις και δίνω το λόγο στον ε, ε, κύριο Μπούλμαν. Ευχαριστώ κύριε Μόντι. Πολύ μου άρεσε η εισαγωγή σας. Και εντωμεταξύ Έχετε γερμανική μετάφραση. Ωραία. Λοιπόν, πολύ μου άρεσε η, η εισαγωγή σας. Ήταν ε, πολύ έξυπνη. Μου άρεσε και ο παραλληλισμός με το 2003 και η σε αλληλεπιδράσεις ε, μεταξύ των ε, διαφόρων εμπλεκομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίοι προσιλώνονται εις ε, τις βραχυπρόθεσμες προεπτικές και παραβλέπουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο περισσότερο είναι τι σημαίνει αυτή η διαπίστωση για την κατάρταση του πακέτου το οποίο είναι προσυζήτηση. Πού κινδυνεύουμε ε, να ξεχάσουμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, πώς πρέπει να κατευθυνθεί το Κοινοβούλιο κατά τρόπον ώστε να προσαρμοστεί στις ε, και κλικές ε, επιταγές της δημοσιονομικής πολιτικής και πόσο πρέπει κανείς να κινηθεί κατά τρόπον ώστε ε, να λάβουμε υπόψη τις διάφορες οικονομικές δομές των διαφόρων κρατών μελών. Δηλαδή πώς θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και θα τα εντάξουμε εις ε, το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης. Ε, διότι εδώ θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες και να δούμε πώς θα μπορέσουν όλα αυτά να ενταχθούν στις μακροπρόθεσμες προπτικές του πακέτου. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το σχόλιο σας για τα ευρωμόλογα. Είσαστε πιστικός και σαν Γερμανός σας πιστεύω, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να υπάρξει ένας θεσμικός σχεδιασμός για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθούν αυτά τα ευρωμόλογα. Θα ασχοληθεί με αυτά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ορισμένα σχόλια περαιτέρω ε, θα ήταν ευπρόσδεκτα επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, υποθέτω ότι τώρα έχουμε τους μισούς ομιλητές που ζήτησαν το λόγο οπότε κύριε Μόντι ε, θέλετε να σχολιάσετε και να κρατήσετε και λίγο χρόνο για να υπάρξει ένας δεύτερος γύρος. Βέβαια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι. Όσον αφορά τη ρευστότητα και το θέμα που έθεσε η κυρία Φόρντ είναι πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να περιληφθεί και με μεγάλη προσοχή στη συζήτηση. Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις του δημοσίου τομέα με ρωτάτε αν έχω περαιτέρω σκέψεις όσον αφορά την έκφραση με αριθμούς ε, και πώς τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να θα μπορούσαν να περιλάβουν τα πάντα ως επενδύσεις για να παρακάμψουν τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι το 1996 συζητήσαμε για πρώτη φορά το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχα πει τότε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για να καταρτήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά αν ξεκινήσουμε με το Eurostat, με τους οικονομολόγους και καθορίσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για επενδύσεις, σε μερικά χρόνια θα έχουμε προχωρήσει. Και η προσέγγιση αυτή θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο διότι θεωρούσαμε ότι ήταν επικίνδυνο να σκεφτούμε κάτι τέτοιο και θα πρέπει πάντοτε ε, στην οικονομία αλλά και ιδίως στη ζωή να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ της ε, πρώτης ε, ε, τάξεως και της δευτέρας τάξεως. Δηλαδή, καταρχήν το να σκεφτούμε τι είναι η επένδυση είναι μια σημαντική δυσκολία δευτέρας τάξεως. Η πρώτη τάξη είναι αν συμφωνούμε ότι ε, η σωστή ιδιωτική επένδυση ε, με δημόσια εποπτεία είναι καλύτερη από οποιαδήποτε δημόσια επένδυση. Εάν έχουμε πρόβλημα με αυτό ας το εξετάσουμε. Θα πρέπει λοιπόν οι ορισμοί μας να είναι πάρα πολύ περιοριστικοί αρκεί να έχουμε συμφωνήσει ε, για ένα θέμα το οποίο σε γενικές γραμμές ασχολείται με μελλοντικές Επίση, Επίσης, ε, με ρωτήσατε τι έγινε με την εμπειρία του 2003 και τώρα πόσο μπορώ ε, να προβλέψω ή στο κείμενο το οποίο έχετε μπροστά σας περισσότερη δημοσιονομική προσοχή. Εχθές ο πρόεδρος Μπάους προείδρευσε μια συζήτηση όπου πολλοί μίλησαν για το οικονομικό πακέτο χωρίς να αισθάνονται ότι περιορίζονται από το υπάρχον κείμενο και υπήρξαν διάφορες θετικές και ριζικές κριτικές και θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι εσείς γνωρίζεστε βάσει ενός προγράμματος το οποίο είναι έξυπνο, είναι λογικό και είναι μία από τις ε, εφικτές ε, λύσεις. Εφόσον λοιπόν έχετε αυτό το κείμενο, αυτή τη σειρά των κειμένων μάλλον προς επεξεργασία υπάρχουν διάφοροι τρόποι και ε, ε, μία, ένα θέμα το οποίο πρέπει να αποφύγουμε για την αξιόπιστη περι, ε, βραχυπρόθεσμη πειθαρχία είναι όπως λέγεται στο κείμενο να ποσοστοποιήσει κανείς τα κριτήρια για να περιληφθεί ε, το χρέος στο ποσοστό του ΑΕΠ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στο νέο κείμενο αλλά αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι όλα αυτά να γίνουν στα πλαίσια της κοινή λογικής Δηλαδή, εάν θέλει κανείς ε, να ε, καθησυχάσει τη δημόσια γνώμη βραχυπρόθεσμα και πείτε ότι είναι αδύνατον να περιληφθεί αυτό το ποσοστό, τότε ε, είτε δημιουργείται δυσπιστία προς τον ενδιαφερόμενο ή καταστρέφεται και προκαλείται μια κρίση στα οικονομικά της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος επεξεργασίας του κειμένου όπου να εξετάζει κανείς και το θέμα των δημοσίων επενδύσεων. Και ε, για να διασφαλίσετε ότι δεν πρόκειται να διλύσετε την πειθαρχία, εγώ παραδείγματος χάρη θα ήμουν υπέρ μιας μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής τώρα μιλούσαμε ε, για 3% αποκλήσεως από το ΑΕΠ ε, ε, γιατί λοιπόν να έχουμε κάτι τέτοιο ποιος το καθόρισε και όσον αφορά το θεσμικό σχεδιασμό θα σας έλεγα ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα κοινοτικό οργανισμός ο οποίος θα εξέδιδε αυτά τα ευρωμόλογα για να μην πολλαπλασιάσουμε τα, τους διάφορους οργανισμούς και υποθέτω ότι το Κοινοβούλιο είναι πολύ ευαίσθητο στο θέμα αυτό. για το EFSF. Υποθέτω ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Τώρα έχω τέσσερις ομιλητές, οπότε θα σας πάρω σε δύο ομάδες των δύο για να είμαστε πιο δυναμικοί. Πρώτα ο Φίλιπς, μετά η Σιλβή, μετά ο Μάριο και μετά οι δύο επόμενοι ερωτούντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καθηγητά Μόντι για την τοποθέτησή σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον οι ιδέες που μας είπατε. Εσείς αναφέρατε τα δύο είναι Ανδεστισμό, εντεγκρασιό, επενδύσεις και ολοκλήρωση. Μπορούμε να έχουμε εμείς μια πραγματική οικονομική ολοκλήρωση χωρίς να έχουμε αυτό που ο Τρισέ ονομάζει μια φορολογική ομοσπονδία εγώ δεν μιλώ για τη λίγο σχιζοφρενική φορολογική ομοσπονδία του Τρισέ που αφορά μόνο στο κεφάλαιο των δαπανών. Εγώ μιλάω για το κεφάλαιο εσόδων. Εσείς το αναφέρατε στην έκθεσή σας για την εσωτερική αγορά, υπό την οπτική δηλαδή της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού. Ε, ρωτώ, αν δεν έχουμε φορολογικά έσοδα και δεν έχουμε ένα μίνιμουμ συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών μπορούμε να καταλήξουμε σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα μήλο φορολόγηση των επιχειρήσεων κατά πολέμηση της απάτης φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών πράξεων είναι δυνατόν χωρίς όλα αυτά να έχουμε εμεί μία βαθμίδα ολοκλήρωσης για να πετύχουμε την ΟΝΕ και το δεύτερο κεφάλαιο συνδέεται άμεσα με αυτό. Δεν υπάρχει ολοκληρώση αν δεν έχουμε κοινά σχέδια. Κοινά επενδυτικά σχέδια, ας πούμε, στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και επενδύσεις όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι μέσα που μέσα από την ίδια τους την δυναμική κοινών σχεδίων μπορούν να οδηγήσουν σε ολοκλήρωση. Εσείς τι σκέφτεστε για όλα αυτά. Σιλβί. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά που είστε εδώ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για αυτά που είπατε για το Κοινοβούλιο και για, αυτά, και για τις εργασίες του, αλλά για το γεγονός ότι καταλάβατε υπό ποιο πνεύμα εργαζόμαστε. Από έξω πολλοί κόσμος ε, <coughs> σχηματοποιεί σαν καρικατούρα το, τη δουλειά του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορέσατε να καταλάβετε όλο αυτό το ζήτημα της διαφάνειας. Πρόκειται για, μια σχέση, ε, για ένα θέμα που δημιουργεί περίεργες ε, σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, είναι ένα σημείο λοιπόν πολύ σημαντικό. Το ίδιο και για τα ευρωομόλογα. Σας ευχαριστώ που επιμείνατε στα στοιχεία εκείνα που μπορούν να πείσουν τις χώρες που είναι ιδιαίτερα δεμένες με το θέμα της πειθαρχία. Το λέω και εγώ στην έκθεσή μου, όχι για να διευκολύνουμε μία ανεύθυνη συμπεριφορά, αλλά για να ξαναβρούμε την πειθαρχία της αγοράς. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό το οποίο είπατε το 96 έχει δημοσιευθεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως να γίνει κάτι τέτοιο γιατί καλές ιδέες χρειάζονται χρόνο για να προχωρήσουν. Αν μας δίνατε λοιπόν μερικές αναφορές, ε, εγώ πραγματικά θα τις ήθελα. Και δεύτερον είναι η πολύ τεκμηριωμένη παρατήρηση που κάνατε και παραπέμπει στην έκθεσή σας στον παγκόσμιο χαρακτήρα της οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν μπορούμε εμείς να ενισχύσουμε την ΟΝΕ χωρίς να έχουμε κάνει κάτι και στον τομέα αυτό. Πώς μπορούμε να ξαναβρούμε αυτήν τη συνοχή. Δεν μπορούμε εμείς να εντάξουμε το Single Market Act στο πακέτο μας. Όμως και τα δύο πρέπει να τα εξετάζουμε από κοινού. Πώς μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μία διασύνδεση μεταξύ των δύο. Και εγώ στην έκθεσή μου προχωρώ πολύ μακρύτερα από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Τι μπορούμε λοιπόν να βάλουμε εμείς πιο συγκεκριμένα σε αυτό το πακέτο Euh, Κύριε Λαμπέρ, η απάντησή μου είναι ναι σε όλες σας τις ερωτήσεις. Δηλαδή, πιστεύω όπως και εσείς ότι δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορούμε να έχουμε μια πραγματική οικονομική ολοκλήρωση χωρίς να υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο στη φορολόγηση και κοινά επενδυτικά σχέδια για την φορολόγηση και από αυτήν την πλευρά και για την κοινή μοίρα δηλαδή της Ευρώπης δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε χρειάζεται μάλλον να πειράξουμε το θέμα των ιδίων πόρων ή τα θέματα των τίτλων ε, στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι κατά, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα άλλο θέμα. Δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε, ότι θα χρειαζόταν μία φορολογική ομοσπονδία για να έχουμε μία αηφόρο ή ο ναι. Διότι όταν μιλάμε εμείς για τον όρο φυσκάλ φορολογικό, τι είναι, είναι δημοσιονομικό, είναι θέμα εσόδων, τι είναι. διότι από δημοσιονομικής πλευράς ο μηχανισμός που έχουμε μπροστά μας αποτελεί πρόοδο. Και πιστεύω, όπως και εσείς, ότι είναι απόλυτα απαραίτητη ε, ένας συντονισμός των φορολογικών συστημάτων για να λειτουργήσει μια ενιαία αγορά και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε ένα συγκεκριμένο τομέα ε, σε συγκεκριμένου, συγγνώμη, τομείς της φορολόγησης. Μερικά θέματα είναι ταμπού. Διότι όλοι συμφωνούμε τελικά ότι είναι ταμπού και γι' αυτό πρέπει να τα θεωρήσουμε ταμπού. Και αυτό είναι καταστροφικό. Στον φορολογικό συντονισμό μπορούμε να προχωρήσουμε. Το 97 εμείς κάναμε το πρώτο μικρό φορολογικό πακέτο με τον κώδικα και όλες για την καλή συμπεριφορά των ε, επιχειρήσεων κλπ. Και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε όμως σήμερα εμείς να μιλάμε. Σήμερα το έγραψα εξάλλου και στην έκθεσή μου ε, και ανέφερα ως πρώτο μέτρο softly softly γλυκά γλυκά η ομάδα φορολογικής πολιτικής να αναστηθεί. Και αναστήθηκε. Ήταν το μέσο που χρησιμοποίησαμε για το πρώτο φορολογικό πακέτο. Και το είχαν ζητήσει το Συμβούλιο Υπουργών που είναι πιο πολιτικό όργανο και όχι Κορεπέρ. Και προεδρεύεται αυτή η Επιτροπή σήμερα, ε, είναι στη δεύτερη συνεδρίαση, προεδρεύεται από τον Επίτροπο Σεμέτα και αποτελεί δηλαδή ένα χώρο προβληματισμού και σκέψης. Σύμφωνο λοιπόν μαζί σας ότι δεν πρέπει να είμαστε απόλυτα απεσιόδοξοι και για τα σχέδια κοινών επενδύσεων και εδώ σύμφωνο απόλυτα όλοι εργαζόμαστε για τη δημιουργία της ενιαίας νομοθετικής αγοράς. Χρειάζεται όμως και η φυσική αγορά, η απτή αγορά. Διότι αλλιώς η εσωτερική αγορά στο σύνολό της δεν θα λειτουργήσει. Δεν είναι πλέον ευτυχείς οι πολίτες και η πολιτική υποστήριξη δεν είναι πλέον ε, ορατή. Κυρία Αγκουλάχ, σας ευχαριστώ που αναφέρατε ότι κατάλαβα αυτό που θέλετε εσείς να πείτε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προχωρήσω λίγο μακρύτερα και να πω το εξής. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό το ότι κατάλαβα αλλά αυτός δεν είναι ο τελικός σας στόχος. για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι απλά και μόνο ένα ευγενές ε, όργανο το κοινοβούλιο αλλά όμως και συντεχνιακό ταυτόχρονα. Θα πρέπει να πληρώσουμε ένα τίμημα δημοσιονομικής απειθαρχίας για να δώσουμε αυτόν τον πιο ανοιχτό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορατότητα προς τους πολίτες. Δεν πιστεύω. Ξέρετε ότι σε όλες τις χώρες έχουμε θέση ε, κάποιους φραγμούς στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών κοινοβουλίων. Ε, βέβαια στη δική σας περίπτωση τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά για τα ευρωμόλογα. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που είπατε για τις δύο τώρα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Βεβαίω να σας δώσω τα στοιχεία. Η θέση του 96 είναι δημόσια θέση διότι και σε αυτήν την προϊστορική περίοδο ε, υπήρχαν τα σχετικά ΜΜΕ και συζητήθηκε η επιστολή που είχα στείλει στον πρόεδρο της Κομισιόν επαρκώς στον τύπο. Α, και ποια ήταν η άλλη ερώτηση, η σχέση, ο δεσμός με, το, με τη single market. αν μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών θέλετε να αναφερόμαστε όχι μόνο σε αυτές που αφορούν στα κράτη-μέλη, διότι εμείς αξιολογούμε τη δική τους μεμονωμένη θέση, αλλά θέλετε να αξιολογούμε την συλλογικά τη διαρθρωτική πολιτική της Ένωσης τότε μπορούμε κάλλιστα να εντάξουμε και την εσωτερική αγορά. Και μπορείτε μάλιστα να επιχειρηματολογήσετε και με το επιχείρημα που αρέσει ιδιαίτερα στον πρόεδρο Τρισέ. Δηλαδή ότι για να έχουμε ένα optimum ΩΝΕ, ναι, μία νομισματική ζώνη που έχει πιθανότητες επιβίωσης θα έλεγα εγώ, θα πρέπει να καλύπτεται από ε, πραγματική ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, το 1996 θυμάμαι ότι υπήρξαν ορισμένα σχόλια όταν ξεκινούσε η Ευρωζώνη και θεώρησα ότι υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να είναι πιο εκτενή και ενδεχομένως και πιο δαπανηρά όταν χρειαζόταν επιδιορθώσουμε κάτι αντί να ξεκινήσουμε κάτι νέο. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε δειλοί στα μέτρα που θα λάβουμε τώρα διότι αν δεν επαρκέσουν θα χρειαστούν επισκευές και αύξηση συνεχής των εξόδων. Έχω ακόμη τρεις ομιλητές, τον Γιούργεν ε, και μετά άλλους δύο ομιλητές που θέλουν να παρέμφουν. Ευχαριστώ σας και ευχαριστώ τον πρόεδρο Μόντι για την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή του, ομιλία του. Μας παρουσίασε τις διάφορες ε, σκέψεις που θα μπορούσαν να μας καθοδηγήσουν για τις συζητήσεις μας στο μέλλον. Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες ερωτήσεις και ταυτόχρονα να πω ότι ήδη είμαστε σε μια επιτυχημένη διαδικασία για έξι εκθέσεις σχετικές με την οικονομική διακυβέρνηση. Ο κύριος Μόντι αναφέρθηκε σε δύο ελλείψεις της διαδικασίας. Η πρώτη αφορά την πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη αγορά, η άλλη αφορά τις ε, επενδύσεις, τις δαπάνες, επενδύσεων, τις επενδυτικές δαπάνες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να ρωτήσω και είναι εγωιστικό σχετικά με το πακέτο αυτό θα ήταν ποια συμπληρώματα θα απαιτούσε, ποια μέτρα θα απαιτούσε η ολοκλήρωση των αγορών κατά την άποψή του. Και επίσης η κριτική σχετική με τις δαπάνες. Πιστεύετε ότι θα πρέπει η διάκριση να μην είναι ε, μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών δαπανών αλλά μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, δηλαδή επενδυτικών δαπανών. Και αν μιλάμε για επενδυτικές δαπάνες, θα παρατηρούν να υπάρχει σχετική πειθαρχία. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη χώρα μου την Πορτογαλία είναι δυνατόν κανείς να ταξιδέψει στον αυτοκινητόδρομο να ταξιδέψει από την ε, πρωτεύουσα στην συμπρωτεύουσα ε, με τρεις διαφορετικούς αυτοκινητοδρόμους παράλληλους έναν τον άλλον και έχουμε αυτοκινητοδρόμους όπου ο ένας ε, έχει πάρα πολύ κίνηση και άλλοι δύο όχι και αυτό γιατί διότι ο καθένας, κάθε πολίτης θέλει να έχει έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο σπίτι του πώς μπορούμε εμείς να, ε, να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταστρατηγήσουμε τις ε, επενδύσεις υποδομών σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερο, ο Επίτροπος ε, άσκησε κριτική για τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού. Υπογράμμισε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί σίγουρα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο αλλαγή των επιλογών αλλά η επιλογή, η δημοσιονομική πειθαρχία δηλαδή, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, διότι τα κράτη είναι αυτά που παρουσιάζουν τον προϋπολογισμό και έχουν πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τις δημοσιονομικές τους επιλογές. Ένας τρόπος λοιπόν για να πειθαρχήσει κανείς ε, τις κυβερνήσεις είναι να υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτως ώστε να χρησιμοποιείται αυτό το δίκτυο ως, ως μέσο πειθαρχίας. Ευχαριστώ. Βλέπω <clears throat> ότι έχουμε πίεση χρόνου, πρέπει να βιαζόμαστε λίγο για να προχωρήσουμε και να προλάβουν όλοι να μιλήσουν. Άστριτ, Λούλινγκ. <laughs> Euh, euh, euh, λοιπόν, <coughs> ευχαριστώ κύριε Μόντε για τις εξηγήσεις, αφέστατες εξηγήσεις ως ήθιστε. για αυτά που είπατε για τις δραματικές επιπτώσεις ορισμένων καταστρεπτικών δηλώσεων ορισμένων κυβερνήσεων αλλά δεν είναι μόνο οι καταστροφικές και καταστρεπτικές ε, δηλώσεις των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων αλλά και του Προέδρου της Επιτροπής όπως άκουσα εγώ σήμερα το πρωί στη γερμανική τηλεόραση. Λοιπόν για τα θέματα πειθαρχία. πιστεύετε εσείς κύριε Μούντι ότι τέτοιες σοφιστικέ, τέτοιες δηλαδή πολύπλοκες διαδικασίες και τέτοιοι αυτοματισμοί μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη-μέλη ή πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Πιστεύετε εσείς ότι τα κράτη-μέλη κατάλαβαν και καταλαβαίνουν πάντα ε, το τι απαιτεί ή ο ναι δεν αποτελεί ψευδέστηση το να πιστεύουμε εμείς σε μία δημοσιονομική πειθαρχία όταν τα κράτη-μέλη δεν έχουν απόλυτη συνέστηση ή συνείδηση καλύτερα της πρόκλησης. Τώρα για αυτό το περίφημο ευρωπαϊκό εξάμεινο όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά όταν βλέπω εγώ ότι στη χώρα μου έχουν μπει πίσω από το δοφράγματα τα, τα συνδικάτα κατά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δεν ξέρω αν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το ρόλο του. Για τα ευρωομόλογα. Είπατε ότι τα ευρωομόλογα, άμα κατάλαβα καλά, θα πρέπει να αποτελούν ένα μέσο διαχείρισης του χρέους όχι ένα μέσο για τις μεγάλες επενδύσεις, για τα μεγάλα ευρωπαϊκά σχέδια. Γιατί. Γιατί εσείς δεν ε, θεωρείτε ότι τα ορφρομόλογα μπορεί να αποτελέσουν ένα μέσο επενδύσεων, ε, μεγάλων επενδύσεων, για παράδειγμα μεγάλα διαρθρωτικά, ε, διαρθρωτικές επενδύσεις. Τώρα για την ενιαία αγορά, πιο ολοκληρωμένη η ενιαία αγορά, εσείς μιλήσατε για φορολογικό συντονισμό, φορολογική ομοσπονδία. Δεν φτάνει όμως αυτό. Χρειάζεται και ένα συντονισμό σε ελαχίστων κανόνων σε όλα τα επίπεδα. Ας πούμε το κοινωνικό ντάμπινγκ, το οποίο υφίσταται ακόμα μεταξύ κρατών μελών. Στην ε, Γερμανία λέμε ότι έχουμε 800 ευρώ κατώτερο μισθό στο Λουξεμβούργο για τους ανειδίκευτους είναι 1800 ε, και ακόμη παραπάνω για τους ειδικευμένους και εδώ κάτι θα έπρεπε να γίνει. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μόνκη, κύριε Μόνκη, κύριε Καθηγητά, Αναφερθήκατε στην έκθεση σας για την ε, εσωτερική αγορά και τις σχέσεις μεταξύ της οικονομικής διακυβέρνησης και της περαιτέρω ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Πριν όμως ο τύπος λέει και επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρεμβαίνει ιδιαίτερος ε, υπέρ των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση του ευρώ και δεν κάνει αρκετά για την ολοκλήρωση της εσωτερικής οικονομικής αγοράς. Φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρές βέβαια οι προτάσεις σας μέσα στην εκθέση, αλλά τελικά οι προθέσεις δεν αρκούσαν για να αλλάξουν συμπεριφορές. Ένα άλλο πράγμα το οποίο ε, επίσης και εσείς δείξατε είναι καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των μακροοικονομικών ρυθμίσεων στην αγορά του ευρώ και η ολοκλήρωση της εταιρικής αγοράς. Στα δύο αυτά καθήκοντα ε, η Επιτροπή επέλεξε να ε, αναθέσει διαφορετικά χαρτοφυλάκια σε δύο διαφορετικούς επιτρόπους. Γιατί θα υπάρχουν δύο διαφορετικές επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε εσείς να εντοπίσετε το σημείο της καλύτερης συνεργασίας, ώστε κατά τον ιδανικότερο τρόπο να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ευχαριστώ. Ε, έλα και στην αλλά σύντομα σε παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε, βλέπω μόνο τρεις βουλευτές που ήταν παρόντες όταν αναλάβατε για πρώτη φορά καθήκοντα επιτρόπου το 94 με 99. Πάντως εμείς οι παλιοί σας θυμόμαστε και εκτιμούμε πολύ τη δουλειά σας. Για τα κριτήρια του Μαστρίχτ. Το 60% ως όριο έγινε δεκτό από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ως κριτήριο του ε, το 30%, το 3% κ. για το νέο χρέος είχε στηριχθεί στο 10%, στο 10% του Τη χρέωση του προηγούμενου έτου. Και με βάση αυτό έγινε ο υπολογισμό όπου υπόθηκε ότι το 3% πρέπει να το μέχρι στο νέο χρέο. Δεν ήταν δηλαδή όπως μερικές φορές ε, ακούγεται αυθαίρετη επιλογή απλώς λεγόταν ότι δεν πρέπει να υπάρχει νέο χρέος, δεν πρέπει να υπάρξει νέο χρέος και αν υπάρξει μέχρι 3% το πολύ. Λέτε ότι η μεγάλη αμαρτωλή στην αρχή ήταν η Γερμανία και η Γαλλία και εσείς ως ε, αρμόδιος επιτροπός τότε είχατε μιλήσει και με τον Επίτροπο για, την, ε, για τον ανταγωνισμό και είχατε προχωρήσει σε προσφυγή κατά των δύο κρατών και έτσι άλλαξε αντίστοιχα και η διατύπωση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη το 2005 για να γίνουν πιο σαφεί και οξύσιοι οι όροι. Ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω, διότι χωρί τροποποίηση τη συνθήκη και ειδικότερα του άρθρου 125 δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτή η εξέλιξη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι άποψη έχετε γι' αυτό. Δεύτερον, για την παρατήρηση σα για την ε, Γερμανία και τα γνωρίζουν πολύ καλά ο κύριο Μπούλμαν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχει απόφαση του ε, Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία δεσμεύει τη γερμανική κυβέρνηση, δεν μπορεί να, παραβιάσει απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και φαντάζεστε ότι αυτό είναι δεδομένο. Είναι άλλωστε παράδοση μεγάλη μακριά στην Γερμανία. Επίσης ε, για την ε, για το μέτρο διάσωση το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μπαρόσο. Ναι, μπορεί να είναι ο πρώτος, είναι όμω και υπεύθυνο ε, για αυτές τις αποφάσεις, αλλά το πιο σημαντικό που θέλω να επισημάνω από τις δηλώσεις Μπαρόσο είναι ότι είπε ότι στο μέλλον το μόνο ε, βαρύνων στοιχείο θα είναι οι προϋποθέσεις του συμφώνου του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη του Μάστρικ. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν ω κριτήρια η επιπλέον επιβάρυνση, τα επιπλέον επιτόκια κτλ. Αυτά από τι τεσσινέ παρατηρήσεις του κ. Μπαρόσου. Και υπενθυμίζω ότι πλέον δεν σας βλέπουμε ως επίτροπο, αλλά ως έναν αντικειμενικό, ειδικό, επαΐοντα και αντίστοιχα εκτιμούμε βεβαίω και, την κρίση σας. Κυρία Μπόουλς, ε, βέβαια τώρα έχουμε ροκανίσει το χρόνο μας, θα πρέπει να είμαστε στο δυνατόν πιο σύντομοι. Αλλά βέβαια οι παρατηρήσεις προξενούν πάλι πολλές απαντήσεις. Κύριο Σμόντσι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει το πιο σημαντικό κομμάτι της ε, συζήτησης και το πιο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν θέλω να φάω το χρόνο των άλλων ομιλητών που περιμένουν. Θα ζητήσω συγγνώμη από τους ε, κυρίες και κυρίους βουλευτές, γιατί θα είμαι πολύ σύντομο τώρα. Τον κύριο Φέιο, τα συγκεκριμένα μέτρα ολοκλήρωση των αγορών. Πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι σας, και βέβαια και εμένα θα πρέπει να με απασχολήσει αυτό, να κοιτάξετε όχι τα συγκεκριμένα μέτρα, γιατί υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις στην πρόταση της, ενίας, της πράξης την ενιαία αγορά του κυρίου Μπαρνιέ, αλλά να βρείτε τη διόρυγα που θα σας περάσει μετα, από αυτήν την πράξη σε μια πιο ουσιαστική και αποτελεσματική λύση για τη διακυβέρνηση. Επίσης, για να πατήσω στον κύριο Σφάπ και να συμπληρώσω κάτι που λησμόνισα δηλαδή ε, στην απάντησή μου για την κυρία Κουλάρ, πώς μπορεί να διασυνδεθεί η δέσμη μέτρων για τη διακυβέρνηση με την εσωτερική αγορά, στην οποία ξέρουμε ε, ε, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο κ. Σφάπ. Και γιατί δεν μπορούσε να προταθεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό, ένα συμβούλιο υπουργών οικονομικών ε, να ασχοληθεί ειδικά με τα θέματα της εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή να τονίσει πάνω απ' όλα ε, όχι απλώ ότι χρειάζεται μια εσωτερική αγορά, αλλά να προχωρήσει και αυτό σε επίπεδο συνόδου κορυφή σημαίνει ότι θα πρέπει οι πρωθυπουργοί, οι αρχή κράτων και κυβερνήσεων να κάνουν ένα συμβούλιο από το οποίο θα προκύψει ότι κάνουν ό,τι μπορούν για την καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση της ε, Ευρώπης. Πάνω από όλο αυτό το, το συμβολικό χαρακτήρα δηλαδή. Ίσως θα μπορούσε να προτείνει κάτι σχετικό το Κοινοβούλιο. Για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις η παρατήρηση σχετική με του τρει διαφορετικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέουν τι δύο ίδιε πορτογαλικέ πόλει είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ασφαλώ δεν προάγει ιδιαίτερα την ιδέα των δημοσίων επενδύσεων, ότι θα πρέπει να υπάρχουν δημοσίε επενδύσει, αλλά από την άλλη πιστεύουμε, φαντάζομαι όλοι, ότι τα εθνικά πολιτικά συστήματα είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε, και αυτό συνήθω επιτελούν, κατά τρόπον ώστε ο πολίτης ε, να είναι σε θέση να ελέγχει το τι πράττει το κράτος ε, με τα φορολογικά έσοδα. Κάποιου τύπου έλεγχος, κάποιου τύπου συνέπειες υπάρχουν. Η άλλη παρατήρηση του κ. Φέγιο. Ναι, θεωρώ ότι είναι πιθανόν και καλό να διανοηθούμε την συστασία ενός ε, δικτύου μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ευαισθητοποιεί τα Εθνικά Κοινοβούλια ω προ την Ευρωπαϊκή Διάσταση των θεμάτων που έχουν να συστήσουν, Για την κυρία Λούλινγκ. Με εύστοχες παρατηρήσεις παρενέβη η κυρία Λούλινγκ, όπως πάντα. Μα οι εξεζητημένες διαδικασίες, οι σοφιστικές διαδικασίες επαρκούν ε, για να επιβάλλουν ε, την πειθαρχία όταν τα κράτη δεν έχουν συνέστηση του πράγματος. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιονομικές ε, πειθαρχίες δεν αγνοούνται και έχουμε αρχίσει και αφήνουμε και παράμερα την υπερβολική αυροφροσύνη έναντι των κρατών που δεν λειτουργούν εύρυθμα. Τώρα κυρία μου, θα μπορούσατε να ενθαρρύνετε τον, να εμψυχώσετε τον Λουξεμβούργιο Πρωθυπουργό για να αλλάξει το θεώρημα Γιούνκερ σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία όταν είπε δηλαδή την περίφημη φράση γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε Αλλά πέστε μας πώς να το κάνουμε και μετά να κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτό το επαναλαμβάνει ο καθένας. Ως ε, πεμπτουσία μιας πολιτικής δήλωσης ε, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι η άσκηση καλών πολιτικών δεν οδήγησε ε, σε χάσιμο εκλογών και καλύτερη διάψευση της θέσεως Γιούνκερ είναι ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ, διότι έκανε ένα σωρό μεταρρυθμίσεις στο Λουξεμβούργο, όχι αρκετές, λέει η κυρία Λούλινγκ, ναι αλλά αυτή είναι η θεωρία Λούλινγκ λέει ο κύριος ε, Μόντι και ήδη έκανε αρκετά πράγματα και δεν τον ε, μετά από 16 χρόνια δηλαδή δεν τον ξεπέταξαν οι Λουξεμβουργιανοί πολίτες για τα ευρωμόλογα σας ευχαριστώ που αναφέρατε αυτό το σημείο. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα ήθελα να έχω ευρωμόλογα ως μέσο χρηματοδότησης των επενδύσεων. Εγώ απλώς λέω ότι η συζήτηση για τα ευρωμόλογα έτσι όπως τα συζητάμε εδώ είναι άλλο πράγμα ως, ως μέσο χρηματοδότησης του δημοσίου χρέους. Τώρα για τον κύριο Σβάμπα. Νομίζω και θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν ε, για την ε, ε, εύγλωτη διατύπωση της προοπτικής. Θυμάμαι την συζήτησή μας για τις δημόσιες προμήθειες. Στο μέλλον αδρυμό. Και θυμάμαι πολύ καλά και τα όρια του 60% για το Μάστρικ και τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν. Τις δηλώσεις βαρός ομολογώ δεν τις έχω δει και δεν μπορώ να τις σχολιάσω. Βέβαια μου κεντρήσατε την περιέργεια και θα αναζητήσω το σχετικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που ήμουν τόσο σύντομος σε αυτό τον γύρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. ως συνήθως, όσο πιο πολύ σας βλέπουμε, τόσο πιο πολλές ιδέες γεννιούνται και θέλουμε πιο πολύ να συζητήσουμε μέσα. Δεν θα αργήσουμε φαντάζομαι να βρούμε άλλη μια δικαιολογία για να σας ε, ξανακαλέσουμε εδώ. Άλλωστε πολλοί από εμά σας βλέπουν και ιδιωτικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που είστε εδώ. Και τώρα περνούμε στην ε, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Παρακαλώ τους ομιλητές να λάβουν το λόγο να έρθουν μάλλον στο Προεδρείο ένα πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα, μια διακοπή μάλλον για να οργανωθούμε. Um, <coughs> oh uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και τώρα ε, ζητώ συγγνώμη από τους εμπειρογνώμονες γιατί ως συνήθως ε, αργήσαμε να ξεκινήσουμε και αυτή η καθυστέρηση συνεχίζεται και τώρα προχωράω χωρίς ε, καμία εισαγωγή και θα έχουμε τρεις δεκάλεπτες παρουσιάσεις εκ των οποίων η πρώτη είναι από τον Paul de ο οποίος είναι καθηγητής ε, διεθνών οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λέβεν. Ε, um, θα ήθελα στην ομιλία μου να ασχοληθώ με τα ευρωομόλογα και δεδομένου του περιορισμένου χρόνου θα ήθελα να ασχοληθώ με τα ευρωομόλογα και το, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Διότι ξέρετε ότι η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει μία υπαρξιακή κρίση η οποία είχε το καλό αποτέλεσμα να βελτιώσει την ε, συνένεση ε, ότι χρειάζεται η πολιτική ένωση για να διατηρηθεί η Ευρωζώνη. Αλλά χρειάζεται και η βούληση να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση και η μόνη στρατηγική που έχει παραμείνει είναι μια στρατηγική μικρών βημάτων προς μια πολιτική ένωση. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι θεωρώ ότι το κοινό ομόλογο είναι ένα καλό πρώτο βρήμα για μια πολιτική ενωσή η οποία μπορεί να καθησυχάσει τις χρηματαγορές και να βελτιώσει την κατάσταση της Ευρωζώνης συγχρόνως στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Το βασικό μου επιχείρημα για το κοινό ευρωμόλογο είναι, το, είναι πολιτικό και είναι το εξής. Δηλαδή η κρίση αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη έχει εκφυλιστεί σε μια υπαρξιακή κρίση και πολλοί αναρωτιούνται εάν η Ευρωζώνη όπως την ξέρουμε σήμερα θα επιβιώσει. Η έλλειψη αυτή η εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ευρωζώνης οδηγεί σε ενδημική αστάθεια και μετατρέπει τα κακά νέα για κάποια χώρα σε κακά νέα και για άλλες χώρες με αποτέλεσμα να κινδυνεύει όλο το σύστημα. Η κρίση έχει επιδεινωθεί από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου και ε, του Δεκεμβρίου να πληρώσουν οι κρατούντες τα ευρωομόλογα ε, εάν ε, βοηθηθούν και δημιουργείται μία ανασφάλεια σχετικά με τη φορολογία. Όσον αφορά το ε, ε, ε, διεθνές ε, οικονομικό σύστημα ε, όλοι ήξεραν ότι παρόλο που υπήρχε μία σταθερή ισοτιμία μπορούσαν να υποτιμήσουν το νόμισμά τους και όταν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος είναι προφανές ότι όλοι θεωρούσαν ότι θα υπήρχε υποτίμηση. Το ίδιο γίνεται τώρα στην Ευρωζώνη. Εάν πούμε ότι οι χώρες μπορούν να υποβαθμίσουν τα ομόλογα τους, κάθε φορά που υπάρχει η υποψία ότι ε, κάποιος θα πουλήσει τα ομόλογά του, δίνουν ένα κίνητρο στις κυβερνήσεις να υποτιμήσουν τα ομόλογα τους. Οπότε έτσι έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα πρόβλημα αντί να επιληθεί το πρόβλημα της Ευρωζώνης το οποίο πλέον καθίσταται ενδυμικό και υπαρξιακό. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα αυτό δηλαδή να ξεχάσουμε τις ιδέες να εξασφαλίσουμε ε, όσους έχουν ε, ομόλογα ε, αλλά η δικιά μου γνώμη είναι ότι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο είναι να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα δείξουν στις αγορές ότι ε, σέβονται τις υποχρεώσεις που έχουν λάβει έναντι της Ευρωζώνης. Μέχρι στιγμής έχουμε δηλώσεις οι οποίες δεν είναι παρκείς και αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα δώσει στις αγορές το σήμα ότι οι κυβερνήσεις στηρίζουν την Ευρωζώνη και το κοινό ευρωομόλογο είναι ένας τέτοιος μηχανισμός εκδίδοντας ένα ευρωομόλογο η χώρες ε, θα δείξουν ότι είναι αξιόπιστες ε, για τα μέτρα που έχουν λάβει από κοινού και θα είναι μία δέσμευση που θα πει στις αγορές ότι οι χώρες ε, πιστεύουν στο μέλλον της Ευρωζώνης. Είναι ένας μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο οι κυβερνήσεις δένουν μόνες τους τα χέρια τους και δείχνουν στις αγορές ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια, στο ίδιο καράβι, στην ίδια θέση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η λύση είναι πολιτική και το πρώτο βήμα για μία πολιτική ένωση. Είναι ένας τρόπος να δημιουργήσετε μία πολιτική ένωση αν δημιουργήσετε ένα μηχανισμό που δείχνει ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε και θα υποχρεώσει τις χώρες να λάβουν συγκεκριμένα μέσα για μία πολιτική ένωση και αφαιρεί τους ε, υπαρξιακούς κινδύνους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη και την αποσταθεροποιούν. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους θα χρειαστεί τα ευρωομόλογα και ο Μάριο Μόντι τα ανέφερε. Πιστεύω δε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν, ένα, σαν μια εγγύηση εάν χρησιμοποιηθούν σοφά. Θα σας πω τώρα ποιες είναι οι αντιρρήσεις στα ευρωμόλογα ευρωομόλογα ε, και ε, η αντίδραση αυτή είναι κατανοητή διότι ε, θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι αντιρρήσεις αυτές. Καταρχήν υπάρχει το, ο ηθικός κίνδυνος διότι το ευρωμόλογο έχει κάποια εξασφάλιση για τα κράτη τα οποία συμμετέχουν διότι θα είναι από κοινού υπεύθυνε για το χρέος και ε, θα πρέπει να αποφύγουν να δημιουργήσουν υπερβολικό χρέος και στις χώρες οι οποίες ε, φοβούνται ότι άλλες χώρες μπορεί να ε, να δράσουν προς τη δημιουργία χρέους δημιουργεί ανασφάλεια και αυτή είναι η μία αντίρρηση η οποία υπάρχει η άλλη αντίρρηση αναφέρεται στο ότι οι χώρες που είναι 3α ε, ε, δηλαδή πολύ αξιόπιστες όπως η Γερμανία φοβούνται ότι θα πληρώσουν περισσότερο συμμετέχοντας σε ένα κλαμπ όπου υπάρχουν και χώρες με χαμηλότερη βαθμολόγηση και άρα και αυτές θα χρειαστεί να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια μπαίνοντας στο κοινό καλάθι με τις άλλες ενώ μόνες τους έχουν μία αξιολόγηση 3α στην αγορά. Ε, γι' αυτό και ε, πρέπει να εξετάσουμε πώς αυτό ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί εις το σχεδιασμό των ευρωμολόγων συνδυάζοντας λοιπόν τις δύο ιδέες οι οποίες υπάρχουν να υπάρχουν τα μπλε και κόκκινα ομόλογα η οποία είναι μια ιδέα που έχει υποβληθεί ότι η συμμετοχή στα μπλε ομόλογα θα είναι το υψηλότερο επίπεδο και όσοι έχουν ε, κάποιο χαμηλότερο επίπεδο ΑΕΠ θα έχουν κόκκινα ομόλογα που θα πληρώνουν μεγαλύτερο επιτόκιο στην αγορά για να μπορέσουν έτσι να επιλύσουν και το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου διότι δημιουργείται μία διαφοροποίηση μεταξύ ε, της ε, οριακής, ε, του οριακού κόστους δανεισμού και του μέσου κόστους δανεισμού. Κρατάτε δηλαδή το μέσο κόστος δανεισμού χαμηλότερο από το οριακό κόστος δανεισμού και διευκολύνεται τις χώρες να ε, ε, φύγουν από τη δυσχερή κατάσταση ενώ όσες το παρακάνουν θα χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερο και θα ήθελα αυτό να το συνδυάσω με ένα άλλο χαρακτηριστικό που ε, διατυπώθηκε σε μία πρόταση που κάνουμε δηλαδή διαφοροποίηση των επιτοκίων μεταξύ ε, μπλε και κόκκινων ομολόγων οι χώρες οι οποίες είναι καλύτερες θα έχουν χαμηλότερο επιτόκιο και αυτό δεν θα ισχύει στο κόκκινο ομόλογο. Θα υπάρχει μία ανακατανομή ώστε οι μπλε χώρες να εξασφαλιστούν ότι δεν θα πληρώσουν περισσότερα από αν εξέδιδαν τα ίδια κρατικά ομόλογά τους. Εγώ έτσι βλέπω πώς μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό των αντιρρήσεων και είναι βασικό να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση αυτή για το λόγο που ανέφερα, δηλαδή τον πολιτικό λόγο, να δώσουμε ένα σήμα στην αγορά ότι όλες αυτές οι χώρες είναι σοβαρές και όντως επιθυμούν να διατηρήσουν το ευρώ ως έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα προχωράμε στον Πάολο Μανάς που είναι καθηγητής μακροοικονομικής και ε, διεθνούς οικονομικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε να αναγνώσω την ομιλία μου για να με καταλάβετε καλύτερα. Θα κάνω μια στομή εισαγωγή. Στη συνέχεια θα δώσω κάποιους, ε, κάποιες ιδέες για βράχη και μέσο πρόθεσμες μεταρρυθμίσεις και στη συνέχεια κάποιες, κάποια σχόλια για πτυχές που έχουν να κάνουν με προτάσεις για το Σύμφωνο στο και Ανάπτυξης, ανάπτυξης τη μακροεπιτήρηση και τα άλλα θέματα. Θα σας ε, Ξεκινήσω λοιπόν με την εισαγωγή και ελπίζω ότι το κείμενο θα διανεμηθεί. Ξεκινούμε λοιπόν με την ευρωπαϊκή κρίση δανεισμού χρέους. Ξέρετε ότι τα κρατικά χρέη των πιο ευάλωτων, κρατών μας υπενθυμίζουν διαρκώς Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, ίσως και Ιταλία ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Και αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι ε, οι επενδυτές αναγνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατάλληλους θεσμούς ε, για πρόληψη αλλά και επίλυση κρίσεων. Έχουμε ένα τεράστιο καθήκον λοιπόν μεταρρύθμιση των θεσμών και ίσως δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να το επιτελέσουμε. Οι εθνικέ κυβερνήσει, μερικέ φορές φαίνεται να ανταποκρίνονται μάλλον σε εθνικούς πολιτικούς ε, συσχετισμούς και όχι στο στόχο του κοινού καλού. Σημειώνω δε ότι οι αποφάσει του έχουν, έχουν ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι οι κρίσει, νομισματική, τραπεζική, εταιρική, δημοσίου χρέους, υπενθυμίζουν ότι οι κρίσεις είναι ένα είδος χήμερας, δηλαδή ξεκινούν έρποντας και ξαφνικά αρχίζουν να γιγαντώνονται και ορμάνε πάνω στον θύμα τους. Πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε ότι έχουν ήδη αναλυφθεί ή ανακοινωθεί σημαντικά μέτρα, θέσπιση ενός μόνιμου Ευρωπαϊκού Σταθεροποιητικού Μηχανισμού μετά το 2013 με νέες ρήτρες συλλογική δράσης για, για τη νέα έκδοση ομολόγων, δέσμευση για χρηματοοικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Μέσου δημοσιονομική σταθερότητα μέχρι το 2013, νέε προτάσει για την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, ουσιαστικών προτάσεων μάλλον και για την εφαρμογή ενό νέου πλαισίου μακροοικονομική επιτήρηση, νέα πρόταση για την ανάκαμψη των τραπεζών και την ενίσχυση ομοθεσία και τη επιτήρηση. Πλην όμω τα μέτρα αυτά δεν μπόρεσαν να διασκεδάσουν ανησυχίες σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη πίεση στη χρηματοδότηση, την ε, υποβάθμιση και την, τον κίνδυνο της επιμόλυνσης των γειτονικών οικονομιών. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Είναι μεγάλη κλίμακα μεγέθους για την οποία μιλάμε. Σημαντικό το καθήκον που έχουμε να επιτελέσουμε. Χρειάζεται ως εκ τούτου μια σειρά θεσμικών μεταρρυθμίσεων να αναλυφθεί και η λέξη σειρά έχει κρίσιμη σημασία εδώ καινοτόμες προσεγγίσεις εκεί που απέτυχαν οι παλιές πολιτικές επιλογές. Καταρχάς λοιπόν, βραχή πρόθεσμα για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Πρώτη κατεπίγουσα προτεραιότητα είναι να διευρυνθεί το δανειοληπτικό δυναμικό του EFSF, ESM και να εξασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό αρκετό χρόνο για να προχωρήσουμε στι υπόλοιπε στι μεσοπρόθεσμε δηλαδή μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2,85-3 εκατομμύρια σε δολάρια δάνεια που θα λήξουν την περίοδο 2011-2013. Η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν ε, προθεσμίες στα δάνειά τους ύψους 502 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2011. Άρα χρειάζεται η δανειοδοτική ε, ισχύ του EFSF να ενισχυθεί στο 1,7 με 2-3 εκατομμύρια για να καλύψουν το ενδεχόμενο σωρευτικών ε, ε, ετοιμισμάτων από την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιταλία το 2011-2013. Αυτό μπορεί να γίνει με την επέκταση των δανείων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Ευρωπαϊκό ε, Σύστημα Χρηματοδότηση. Ε, ή την αγορά κρατικών ομολόγων από αυτό, αντί να τα αγοράσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και ούτω καθεξής. Δεύτερο στοιχείο, όπως το ακούστηκε και νωρίτερα, είναι ότι αυτή η δανειοδότης θα πρέπει να είναι μαζική, να, να επιβάλλονται όροι, που, να τη συνοδεύουν όροι και να ε, συνοδεύεται από επιδοτούμενα επιτόκια προκειμένου να διευκολύνει προβλήματα βιωσιμότητας. Επίσης, Χώρε, Μάλλον, θα ήθελα να προβώ μια σημαντική διάκριση μεταξύ των κρατών, οι οποίε παρουσιάζουν προβλήματα ε, ρευστότητα, βραχυπρόθεσμα, και εκείνων που αποδεικνύονται αφαιρέγγυε. Οι αφαιρέγγυε χώρε θα πρέπει μόνο μερό να προβούν σε ένα διάρθρωση του δανείου του το ταχύτερο δυνατό, με την ανταλλαγή προσφορών, όπως είδαμε παραδείγματι στην περίπτωση του Πακιστάν, της Ουκρανίας, της Ουρουγουάης, δεκαετία του 90 η προηγούμενη παρελθούσα εμπειρία ε, ανικανότητας ε, εξυπηρέτησης κρατικών δανείου δείχνει ότι είναι συνήθως περιορισμένο το κόστος που προκύπτει από αυτή την αδυναμία εξυπηρέτησης, περιορισμένο χρονικά και σε όγκο. Άρα χρειάζεται μια σαφής αλλά και διαφανής διάκριση ε, των αφαιρέγγιων χωρών από εκείνες που έχουν πρόβλημα ρευστότητας για να αποφευχθεί η επιμόλυνση της μίας από την άλλη. Ε, επίσης χρειάζεται ε, να έχουμε... Α, έχει τελειώσει ο χρόνος μου, ε. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω να μιλήσω και πιο φυσιολογικά. Μέσω πρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και μετά για τα ευρωομόλογα. Για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Το πρόβλημα κυρίω είναι, πιστεύουμε, η πρόταση ότι η προσαρμογή θα πρέπει να είναι αναλογική ω ε, ως προς το ποσοστό του δανείου επί του ΑΕΠ, το 60% δηλαδή, ε, σε σχέση με το όριο 60% επί του ΑΕΠ. Αυτό όμως, αυτός ο λόγος μπορεί να διγενήσει περισσότερες δυσκολίες. Μπορεί δηλαδή να απαιτεί τα εξή. μπορεί να απαιτεί προσαρμογές μη αξιόπιστε από χώρε υψηλής χρέωση. Φανταστείτε το Βέλιο ή η Ιταλία να προσαρμοστούν να προσαρμόσουν μάλλον ε, το λόγο αυτόν και έτσι το πλεονέκτημα πρωτογενούς ε, ισοζυγίου να ανέλθει στο 4-5% του ΑΕΠ για μια 20 ετία περίπου. Αυτό είναι αναξιόπιστο. Και το θέμα δεν είναι αν ακολουθούμε ή όχι τους κανόνες ή αν ε, ενδεχομένω κιν, σε κίνδυνο επιβολής κυρώσεων όπως βλέπουμε να συμβαίνει για τις περισσότερες χώρες. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα ότι κινδυνεύουμε στην Ευρώπη να έχουμε, δεν το χρειαζόμαστε δηλαδή, δεν θα έπρεπε καθόλου να έχουμε έναν συντονισμένο, μια συντονισμένη φορολογική, δημοσιονομική λιτότητα. Δημοσιονομική λιτότητα η οποία είναι περιττή διότι δεν έχουμε αντίστοιχα οικονομικά δεδομένα στι διάφορε χώρε και ε, ισοσκέληση των προπολογισμών του. Δηλαδή, άλλο θα πρέπει να επιβάλλει περισσότερη, ή λιγότερη λιτότητα και το καθεξή. Από τις προτάσεις που έχουν ακουστεί, Μία που σχετίζεται και με τη δική μου δουλειά λέει ότι θα πρέπει σε αυτόν τον ισχύοντα κανόνα του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη να εισαχθεί, να συμπληρωθεί δηλαδή ένα μηχανισμό αντίστοιχο με αυτόν που κάνουν πολλέ χώρε ε, με το ινάδιο οδηγήσεω. Δηλαδή, αν κάποιο προβεί σε ορισμένε παραβάσει, να χάνει πόντου, να του θερούνται κάποιοι πόντοι και να του ανακτά σιγά σιγά όταν προσαρμόζεται στου κανόνε. Έτσι μπορούν οι χώρες να ε, εισαγάγουν μια πολιτική σταθεροποίησης και ταυτόχρονα να εξασφαλίσετε η απαραίτητη πειθαρχία. Και τώρα θα ήθελα να περάσω σε κάποιους συλλογισμούς για να ολοκληρώσω ως προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χρέους και τα ευρωομόλογα. Όπως και ο πρόεδρος, ο καθηγητής κ. Μόντι και ο κ. Δεγκράου, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια σημεία πολύ σημαντικά. Σε αυτό συμφωνώ. Έχω όμως κάποιες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ως προς τον χρονισμό της εισαγωγής των ευρωομολόγων. Από οικονομικής έποψης, το ομόλογο, κάθε ομόλογο έχει αξία Όσοι του προσδίδει η αγορά με την προσδοκία ότι το πλεόνασμα στο μέλλον θα είναι ικανό να αποπληρώσει το χρέος για το οποίο εκδίδεται το ομόλογο. Ποιος λοιπόν μπορεί να εξασφαλίσει την βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί στο μέλλον. Γιατί επί παραδείγματι ο Γερμανός ή ο Ολλανδός να θέλει να αυξήσει το πλεόνασμά του έτσι ώστε να καλύψει τα ομόλογα, τα ευρωομόλογα και ενδεχομένω αντίστοιχα το χρέος των λεγόμενων μεσογειακών χωρών. Έτσι λοιπόν, εάν δεν υπάρξει πιο σοβαρή, πιο συγκεκριμένη ολοκλήρωση στα δημοσιονομικά και κυρίως κανόνα σχετικός με την δημοσιονομική κυριαρχία των χωρών με σημαντικό έλλειμμα, δεν βλέπω να είναι βιώσιμη η επιλογή αυτή. Για να είναι βιώσιμα τα ευρωομόλογα χρειάζονται πολύ βαθύτερη ολοκλήρωση ως προς τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών. Δεύτερο δύσκολο σημείο της προτάσεις είναι ο χρονισμός. Σας υπενθυμίσω ότι μία πρόταση διαφοροποιεί μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς χρέους. Υπάρχουν ε, διάφοροι τρόποι, δύο διαφορετικοί τρόποι μάλλον το εξετάσουμε αυτό. Πρώτον, ευνηδιαστικά να εισαχθεί αυτή η πρόταση, πράγμα όμως αδύνατο, αν προκειμένου. Δεύτερον, δεύτερος τρόπος να υποβληθεί η πρόταση θα ήταν πρώτα να επιληθεί το πρόβλημα του χρέους, των χωρών που αποδεικνύονται εφερέγγες και μετά να αρχίσει η διατύπωση των προτάσεων εκ του μηδενός. Πλην όμως αυτό σημαίνει ότι δίνεται μια ε, χρονολογία 2013, ένα όριο χρονικό κατά το οποίο θα έχουν επιληθεί τα προβλήματα. Ενώ τώρα κάθε επενδυτής ξέρει ότι αν αγοράσει τώρα πορτογαλικά ομόλογα, στο μέλλον διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει το κεφάλαιό του. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν ένα χρέος τώρα πρωτογενές το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε δεύτερο γενές. Ο κίνδυνος επιδεινώνεται διαρκώς. Ευχαριστώ πολύ, τέλειωσα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε διανύμει το, το κείμενο. Και άρα όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει. Το συγγνώμη από τον κύριο Μανάσε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Και τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Γκούσταφ Χόρν, προκαθηγητή και διευθυντή του Hans Böckler Foundation. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να εξηγήσω λίγο την φιλοσοφία της ε, Οικονομικής Ενώσεως. Τι σημαίνει οικονομικά. Σημαίνει ότι υπάρχει μία συμφωνία να υπάρχει ένα κοινό ποσοστό πλειοθωρισμού το οποίο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακριβώς ε, και λέει ότι πρέπει να είναι ε, στο 2% και είναι ο στόχος τον οποίο κάθε χώρα που συμμετέχει στην Ευρωζώνη πρέπει να σέβεται και να εφαρμόζει στην πολιτική της. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, και να διαπιστώσουμε ότι δεν έχει γίνει σεβαστή στο το ποσοστό αυτό από δύο ομάδες ε, δηλαδή από μία ομάδα χωρών που αφενός είχε πάντοτε υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού από αυτό που είχε καθοριστεί και μία άλλη ομάδα από χώρες που είχε συνεχώς μικρότερο ποσοστό πληθωρισμού. Μπορεί να φαίνεται τεχνικό το θέμα αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις και οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους στην Ευρωζώνη και αυτό δημιουργεί τεράστια ε, διαρθρωτικά ελλείμματα ή στο ισοζύγιο πληρωμών τους και αυξάνει και το εξωτερικό χρέος που δεν είναι μόνο δημόσιο χρέος, ενδέχεται να είναι δημόσιο χρέος αλλά είναι συγχρόνως και ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής αύξηση του εξωτερικού κρέους και οι άλλες χώρες έχοντας συνεχώς πλεονάσματα αυξάνουν το ενεργητικό τους ε, ε, έχοντας ένα πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται περισσότερα. Αλλά αυτή ε, δεν είναι μια βιώσιμη στρατηγική διότι δεν μπορεί κανείς ούτε να χρεώνεται εσαΐ ε, και να εξυπηρετεί τα επιτόκια διότι κάποια στιγμή οι αγορές αντιδρούν και το είδαμε στους τελευταίους μήνες αλλά συγχρόνως ε, υπάρχει και μια επιβάρυνση για τις χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει το χρέος και πρέπει να το διαγράψουν και ε, αυτό είναι η κατάσταση την οποία να αντιμετωπίζει η Γερμανία δηλαδή εκεί θα πρέπει να διαγραφεί διαγραφεί ένα μεγάλο μέρος και δεν ε, καλύπτεται πλέον αυτά στα οποία βασίζονται. Πρέπει λοιπόν ε, να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές και αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό μακροπρόθεσμα και γι' αυτό με τα μεγάλης χαράς βλέπω της προτάσεις ότι υπάρχει ε, μία διαδικασία για υπερβολική αστάθεια η οποία εφαρμόζεται και είναι κάτι που θα πρέπει να εφαρμοστεί όχι υποχρεωτικά στην επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα διότι υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι ε, για τα πλεονάσματα και μπορεί να υπάρχουν και τεχνικοί τεχνικοί λόγοι για τα ελλείμματα αλλά θα πρέπει βάσει των διαπιστώσεων αυτών να διατυπωθεί μία στρατηγική με την οποία να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά ελλείμματα και πλεονάσματα και να τα περιλάβει σε μία πολιτική. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει απλώς να ασχοληθούμε με αυτό το οποίο απετέλεσε τη βάση της συζητήσεως, δηλαδή το δημόσιο ο, χρέος. Στην περίπτωση της Ελλάδας το πρώτο στοιχείο είναι το δημόσιο ο χρέος και αυτό είναι ε, ε, πραγματικό. Πρέπει όμως να δούμε και το χρέο χρέος του ιδιωτικού τομέα και βλέπουμε τις φούσκες οι οποίες αναπτύσσονται στη μία ή την άλλη χώρα και δημιουργούν ε, υπερβολικά ελλείμματα στις τρέχους άμεσες πληρωμές όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Ισπανίας και της Ιρλανδίας. Αυτές οι εξάρτησεις ε, της ε, ε, δομικής, των δομικών χρεών πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα θεσμικό όργανο το οποίο θα αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις και εγώ είμαι υπέρ της αλλαγής που προτείνει το Κοινοβούλιο δηλαδή να δημιουργηθεί ένα τέτοιο θεσμικό όργανο, ονομάστε το όπως θέλετε. Ε, ε, ε, μπορούσε ουσιαστικά να θεωρηθεί ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο κατά τρόπον ώστε να γίνει η ανάλυση των τρεχουσών συναλλαγών που εντοπίζουν τα ελλείμματα και συγχρόνως να μπορέσει να αναπτυχθεί η τεχνική δυνατότητα να προτιταθεί στις χώρες όπου υπάρχει το πρόβλημα ορισμένες πολιτικές, στρατηγικές και λύσεις να επιλύσουν το πρόβλημά τους. Διότι έχει γίνει μια συζήτηση αν έπρεπε κανείς να καλέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην τελευταία κρίση ή όχι. Εμείς χρειάστηκε να απευθυνθούμε σε αυτούς για έναν απλό λόγο, διότι οι τεχνικές δυνατότητες στην Ευρωζώνη δεν υπήρχαν για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των τρεχουσών συναλλαγών. Ε, και αυτό είναι πολιτικό θέμα. Δηλαδή αν χρειάζεστε να τηλεφωνήσετε στη Washington για να λύσετε τα προβλήματά σας ε, βρίσκετε, βρίσκεστε στο ε, G20 δηλαδή το πρόβλημά σας καθίσταται πολιτικό και παγκόσμιο πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς θα έπρεπε να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας και μεταξύ μας γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα τέτοιο τέτοιο όργανο το οποίο θα μας επιτρέψει να επιλύσουμε τα πολιτικά προβλήματα. Και ένα άλλο θέμα ε, το οποίο ε, είναι δύσκολο και έχουν θέσει διάφοροι συναδελφοί είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί το σύστημα αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι τα ευρωομόλογα είναι ο σωστός τρόπος χρηματοδότησης και δεν θα έπρεπε βέβαια να γίνει ανεφόρον. Οι όροι θα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μία πολιτική η οποία θα επιλύσει τα προβλήματα των ανισορροπιών των τρεχουσών συναλλαγών και δεν θα πρέπει να υπάρξει μία ξέφρενη έκδοση τέτοιων ευρωομολόγων, δηλαδή ε, θα πρέπει να είναι κάτω από το 6% του ΑΕΠ, είναι ένας καλός αριθμός για να ξεκινήσουμε ή όπως ελέγχθη ε, θα μπορέσουν να υπάρξουν και δύο κατηγορίες ευρωομολόγων, τα και τα κόκκινα, τα κόκκινα δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με υψηλότερο επιτόκιο. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση θα συμπληρωθεί και ε, θα αποτελέσει μια οικονομική οντότητα διότι αυτή τη στιγμή κατά κάποιον τρόπο είμαστε ατελείς. Έχουμε μια κοινή νομισματική πολιτική αλλά έχουμε αποκλίνουσες φορολογικές πολιτικές οι οποίες δεν μπόρεσαν να καταρτιστούν σωστά για να γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις της νομισματικής ενώσεως. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα θεσμικό όργανο που θα διαπιστώσει και θα παρακολουθεί να μην υπάρξουν λάθη και γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με την ιδέα των ευρωμολόγων. Θα σας πω ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να καταρτιστούν εν ευθέτω χρόνο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, άρα εντωμεταξύ πρέπει να λάβουμε ε, κατεπήγοντα μέτρα και ε, με το ε, διεθνές ε, νομισματικό ταμείο το οποίο θα αντικατασταθεί από μια νέα μορφή ε, θα μπορέσει να επιτρέψει σε χώρες ε, να ε, συμμετάσχουν σε αυτή τη διεργασία και αυτή τη στιγμή βέβαια πρέπει να αποφύγουμε μια πολιτική η οποία είναι αντιφατική και δεν ε, και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επιτόκιο αναχρηματοδοτήσεως το οποίο θα καθορίσει το υπεύθυνο Ινστιτούτο. Ε, και πιστεύω ότι έτσι θα επιτύχουμε τον στόχο μας. Ευχαριστώ. Και τώρα Περνάμε στις ερωτήσεις και θα ήθελα καταρχήν ε, να μας πείτε ποιοι θέλουν να μιλήσουν τώρα ο Ζων Πολ, ο Ιντο και η Περβόνς. Υπάρχει κάποιος άλλος διότι αν δεν ζητήσετε το λόγο τώρα ίσως μην τα παίξω. Ο Ζων Πολ πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τους εισηγητές που παρουσίασαν διευκρινήσεις αλλά αντί για ερωτήσεις ε, θα κάνω ε, ερωτήσεις οι οποίες θα δείξουν ότι εγώ δεν έχω επαρκής γνώσης όσον αφορά τις νομισματικές κινήσεις. Όσον αφορά τις αγορές πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι ικανοποιημένες διότι θέλουν να μετατοπίσουν τον κίνδυνο προς κάποιον άλλον και να μην αναλαμβάνουν κανένα κίνδυνο. Για να μην αναλάβουν κανένα κίνδυνο θα ζητήσουν από τους άλλους να εγγυηθούν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Επίσης μιλάμε για τα ευρωμόλογα, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο ακριβής ορισμός, γιατί ο καθένας που μιλάει για ευρωμόλογα διατυπώνει διαφορετικά αυτό τον όρο. Εάν δηλαδή θα καλυφθεί μέρος του χρέους ή τι. Μεταξύ της αγοράς και της σχιζοφρένειας βλέπω ότι οι αγορές είναι έτοιμες να υπερθεματίσουν τα ομόλογα, τα τα οποία προσφέρει η Ιρλανδία. Δηλαδή ε, ζητάει κάτι κανείς ελπίζοντας ότι θα έχει κάτι παραπάνω και τελικώς ε, ικανοποιούνται με κάτι λιγότερο. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι χώρες να έχουν ε, καλύτερη πολιτική κρίση. Και τελευταία ερώτηση διαπιστώνω ότι καμία χώρα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με λογικούς όρους και είπατε ότι και αυτές χάνουν αλλά όλες μαζί θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν σοβαρά το θέμα είναι ποιος θα αποπληρώσει και πώς. Διότι εγώ εργάστηκα σε μία τράπεζα, υπάρχει το μόνιμο ο, χρέος αλλά κάποια μέρα πρέπει να αποπληρωθούν τα ομόλογα τα οποία κάποιος έχει ε, ε, δώσει και τέλος όσον αφορά την ε, αποπληρωμή του του χρέους θα πρέπει να υπάρξει μία αυστηρή πολιτική για να μπορέσει να αποπληρωθεί το χρέος κάποια μέρα. Θα συγκροτήσω όλες τις ερωτήσεις και δίνω τώρα το λόγο στον Ούντο. Ο κύριος Γκρόβα που μίλησε στην αρχή αναφέρθηκε στις ε, κινήσεις ε, προειδοποίησης και τα σήματα κινδύνου τα οποία προκαλούν πολιτικές δράσεις από νέες προτάσεις κυβερνητικές που επιβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίδραση προκειμένου να αντιμετωπιστεί μόνο και μόνο η κατάσταση. Βλέποντας όμως το πρόβλημα που έχουμε ενώπιον μας, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και όλα αυτά τα οποία συζητούμε, διαπιστώνω ότι απέχουμε πόρο από μια τέτοια ολιστική προσέγγιση, από μια τέτοια γενική θεώρηση και αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλλον χανόμαστε μέσα στι λεπτομέρειες. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Και παραμένουμε παγιδευμένοι στις ιδέες του πρόπερση για το πώς θα πρέπει να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικά τα μέσα που έχουμε, αν δούμε τις προτάσεις της Επιτροπής ως προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Βλέπουμε ότι δεν φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση της πιο ουσιαστικής αντιμετώπισης κατάστασης, μιας γενικότερης ανάλυσης των, ζητημάτων, μιας ευρύτερης προσέγγισης της οικονομικής ε, ρύθμισης και λειτουργίας. Δεν το βλέπω καν. Και ως εκ τούτου, και αυτό ενώ στην καθημερινή μας δουλειά, η συνέπεια θα πρέπει να είναι το πού μπορεί το κοινοβούλιο να αναπτύξει τις αρμοδιότητες, τις δυνατότητες που του προσφέρει το πλέγμα του, ώστε να πιέσει τις άλλα θεσμικά όργανα, κομισιόν και συμβούλιο, ώστε να αποτραπούν οι χειρότερες συνέπειες αυτής της κρίσης. Με αυτό πρέπει να ασχοληθεί το Κοινοβούλιο. Και σε αυτό θα ήθελα να ακούσω κάποιες συμβουλές από κάθε έναν από τους ομιλητές. Ό,τι και να μας πείτε θα ήταν χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη στον καθηγητή Ντεγκρόου γιατί ε, ήρθα μετά την τοποθέτησή του. Αλλά αναφέρατε όμως ε, τα ευρωομόλογα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη. Τι θεωρούν ε, για, την, ε, για τα φορολογικά συστήματα οι προσκεκλημένοι μας, τι θέση τους προσδίδουν Λοιπόν, πώς το εξετάζουν το θέμα, τι θέση του προσδίδουν μέσα στο γενικό πακέτο μεταρρυθμίσεων που συζητάμε. Δεύτερο, στην, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των έξι κειμένων για την οικονομική διακυβέρνηση υπάρχει μία πρωτότυπη αντίληψη που ονομάζεται Prudent Fiscal Policy, σόφρον ε, φορολογική, ε, ε, φορολογική πολιτική. Τι θέλει να πει αυτό το πράγμα. Αντί prudent δεν θα ήταν καλύτερα να λέμε efficient, αποτελεσματική φορολογική πολιτική. Πώς θεωρείτε εσείς, πώς το εξηγείτε το φαινόμενο αυτό της prudent fiscal policy. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σας αναπτύξω εδώ όλο το σκεπτικό, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, το πώς ε, μπορούμε να έχουμε δηλαδή μια φορολογική βάση που θα επιτρέπει μια ανάπτυξη ε, σταθερή και υγιή ε, για να μειώσουμε το χρέος. Εδώ αναφέρετε εσείς όλο το σκεπτικό του κυρίου Ίσινγκ ότι δεν θα πρέπει να μπουν, δεν θα πρέπει να μην προχωρήσουμε σε θεμελιώδεις αλλαγές. Για το θέμα των ευρωομολόγων πρέπει να απαντηθεί άμεσα μια ερώτηση, η ερώτηση συγγνώμη, και για το θέμα δηλαδή της δημιουργίας μιας αγοράς απορρόφησης του χρέους Λοιπόν, πώς εμείς, ποιο θα είναι το ποσοστό, ποιο θα είναι το επιτόκιο για τη χρηματοδότηση αυτού του κυρίαρχου χρέους. Και τελευταίο, Εκεί που λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία προσφυγής επί παραβιάση, λέτε ότι είναι μη ρεαλιστική. Και τίθεται το ζήτημα των δικτών. Εγώ συμμερίζομαι ότι μία προσέγγιση του θέματος καθαρά ποσοτική, χωρίς ποιοτικά στοιχεία, έτσι δηλαδή όπως φαίνεται στην, από την πρόταση της Κομισιόν, δεν πρόκειται να μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, ποιον μηχανισμό εποπτείας μας προτείνεται Πώς οργανώνουμε μία αποτελεσματική διακυβέρνηση δεδομένου ότι μέχρι τώρα οι δείκτες ήταν καθαρά ποσοτικοί δείκτες και όχι ποιοτικοί. Ναι. Τώρα ολοκληρώθηκαν, λοιπόν, οι ερωτήσεις και να ακούσουμε τις απαντήσεις αν την καλοσύνη με τη σειρά για να μην τα μπερδέψουμε και παρακαλώ το πολύ τέσσερα λεπτά για την κάθε απάντηση. Παρακαλώ, ο καθηγητής Δεγκάου, πρώτος. Καταρχήν θα ήθελα να απαντήσω στην ιδιαίτερα εύστοχη ερώτηση του κυρίου Κόζες. Ποιος ξεπληρώνει το χρέος. Μα μία ε, ένα λογικό χρέος, ένα υποφερτό χρέος δεν χρειάζεται να εξοφληθεί. Μπορεί να διατηρηθεί και να επαναχρηματοδοτείται επάπειρον. Πρέπει να δούμε λοιπόν εμείς την αηφορία του χρέους. Αν πρόκειται... Ε, το, το, το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για βάσταχτο χρέος και γι' αυτό τίθεται όλο αυτό το σκεπτικό. Σήμερα η Ιρλανδική κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει 9%. Και οποιοδήποτε χρέος 9% είναι αβάσταχτο. Με 9% και το γερμανικό χρέος είναι αβάσταχτο. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα επιτοκίων. Ένα επιτόκιο το οποίο επέβαλαν οι αγορές, όχι πάντοτε λογικά αυτά τα επιτόκια, το οποίο όμως συνδέονται απόλυτα με τον πανικό. Και μπορούμε τότε σε αυτή τη φάση να κάνουμε άλλα πράγματα. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία δράση που θα οδηγήσει στη μείωση των τόκων του Ιρλανδικού χρέους. Επίσης, το αβάσταχτο ενός χρέους, όπως σας είπα, εξαρτάται από το επιτόκιο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι οι αγορές πέφτουν σε κατάσταση πανικού. Και αυτό, αυτά τα δύο στοιχεία οδηγούν στο αβάσταχτο του χρέους. Και υποστηρίζω εγώ την ιδέα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου, Ευρωπαϊκού Ταμείου που θα μειώσει το άχθος ούτως ώστε αυτή η χώρα να μπορέσει να ξεκινήσει και ένα νέο αναδιορθωτικό πρόγραμμα. Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην παρατήρηση του κυρίου Μπούλμαν, ο οποίος μας κάλεσε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις Εγώ νομίζω ότι αυτό κάνουμε. Είναι το Eurobond μια συγκεκριμένη πρόταση, μία από τις συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι βέβαια η μοναδική, για να προχωρήσουμε. Και ίσως θα ήταν καλό να εξετάσουμε θεσμικές αλλαγές που μπορεί να, αποτελέσουν, να καταστούν απαραίτητες για μια πολιτική ένωση. Όταν ξεκίνησε η Ευρωζώνη θα θυμάστε ότι είχε υποθεί ότι χωρίς πολιτική ένωση δεν θα μπορέσει να επιζήσει η Ευρωζώνη. Ήταν κοινό, κοινός τόπος για τους ε, οικονομολόγους. Ξεκίνησε η Ευρωζώνη ως πολιτικό εγχείρημα και απέτυχε διότι ξεκίνησε χωρίς βήματα προς μια πολιτική ένωση. Τώρα λοιπόν καλούμεθα να προχωρήσουμε πιο προσεκτικά προς μια πολιτική ένωση με βήματα όπως καταρχάς το ευρωομόλογο, δεύτερον ένα ευρωπαϊκό ταμείο ή το συνδυασμό των δύο αυτών και πάντως μέτρα τα οποία θα βεβαιώνουν, θα εξασφαλίζουν, θα αποκλίνουν οι χώρες η μία από την άλλη. Ίσως πάντως θα πρέπει να συμφωνήσω με τον καθηγητή Μανάσε ως προς την ιδέα του δίκτυ. Ο δίκτυς δεν είναι λύση. Δεν πρόκειται ποτέ να δώσει λύσεις. Και το σύμφωνο σταθερότητα είχε στοιχειοθετηθεί πάνω σε μια αντίστοιχη ε, αριθμολογία και δεν επέτυχε. Στις σύγχρονες δημοκρατίες οι πολιτικοί είναι δυνατόν να υποταχθούν στη δύναμη των αριθμών και να εφαρμοστούν αντίστοιχα ε, κυρώσει με βάση του τα αριθμητικά. Επιστημονική φαντασία πολιτική χρειά Μπορεί να είναι αυτό και τίποτε άλλο. Πολιτική δεν είναι να υποτάσσεται κανεί τα νούμερα, είναι να λαμβάνει αποφάσει. Αλλά και πάλι θα έπρεπε εδώ να επισημάνω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να εξασφαλίσουμε πω οι χώρε θα συγκλίνουν και δεν θα ε, κινδυνεύουν να παρασυρθούν σε διαφορετικέ ε, κατευθύνσεις. Όπως είδαμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Καθηγητής Μάνα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ένα ερώτημα από την κυρία Μπερές αφορούσε το νόημα της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και, θα, και οφείλω ασφαλώς εξηγήσεις. Συνετή δημοσιονομική πολιτική εν γέννη σημαίνει πολύ απλά προϋπολογισμό ισοσκελισμένο σε, ένα, σε μια χρήση με ένα μικρό ενδεχομένως έλλειμμα σε μια αρνητική συγκυρία, ε, ένα μικρό πλεόνασμα, αλλά μέσα σε ένα, σε ένα κύκλο επιχειρηματικό πρέπει να υπάρχει ισοσκελισμένος προπολογισμό για, ε, και σταθεροποίηση ε, επί του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει γενικά δηλαδή και δεν είναι τρελή ιδέα. Όπως επεσήμανε και ο Πολ ότι πρέπει να δούμε εάν αυτή η ιδέα είναι βιώσιμη. Για τα ευρωομόλογα και διανούμε ότι δεν είναι ίσως πολύ σαφή τα όσα ακούστηκαν στην παρέμβασή μου, αλλά η αξία ενός ομολόγου σχετίζεται με την υφιστάμενη αξία των πλεονασμάτων που θα το χρηματοδοτήσουν. Ε. Έτσι λοιπόν, εάν εκδοθεί ευρωομόλογο, πρέπει να στηριχθεί αυτό σε ε, έναν υπολογισμό. Ποιο είναι το πλεόνασμα, η μελλοντική αξία δηλαδή που θα έχει αυτό το ευρωομόλογο. Ε, αφού δεν υπάρχει ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα. Αφού είτε έχουμε ευρωπαϊκό προπολογισμό είτε δεν έχουμε. Εάν έχουμε ευρωπαϊκό προπολογισμό, Προφανώς, ε, δεν βλέπω άλλη λύση, οι πλεονασματικές κυβερνήσεις, ε, οι κυβερνήσεις των κρατών που έχουν πλεόνασμα θα χρηματοδοτήσουν αυτό το ομόλογο. Άρα μπορεί πολιτικά να είναι εφικτό το ευρωομόλογο, αλλά μόνο εάν η δημοσιονομική ολοκλήρωση προχωρήσει περαιτέρω και αν αποδεχθούν απώλεια δημοσιονομικής κυριαρχίας οι κυβερνήσεις προ όφελο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργανών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και το επόμενο θέμα για τη χρηματοδότηση. Εγώ είμαι επιφυλακτικό προ την ιδέα ότι το ευρωομόλογο και μόνο θα οδηγήσει σε εξελίξει στη ε, διακυβέρνηση. Γιατί απλούστατα είδαμε και ότι το ενιαίο νόμισμα δεν είχε την ίδια επιτυχία. Δεν οδήγησε δηλαδή σε σύγκληση των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών. Άρα είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε από νομισματικά θέματα. Τα χρήματα για μένα είναι μέσον. Έχω την παραδοσιακή αυτή άποψη. Και αν δεν τα καταφέραμε με το νόμισμα, το ενίο, δεν θα τα καταφέρουμε το ευρωομόλογο. Για δείκτες επιτήρησης. Δεν νομίζω ότι εδώ το ζήτημα είναι αν θα πρέπει να πιστεύουμε στα νούμερα, να τα ακολουθούμε. Δεν νομίζω ότι το έχει κάνει κανείς απιστικά ε, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ούτε νομίζω ότι παίρνει κανείς τα σοβαρά μια τέτοια υπόθεση. Το ερώτημα είναι μόνο ποιοι δείκτες έχουν προταθεί ως κρίσιμοι δείκτες. Αυτοί οι δείκτες λοιπόν ε, τρεχόντων λογαριασμών, παραγωγικότητας κτλ. έχουν σαν στόχο ουσιαστικά να υπάρχει ένα μέτρο για να επιβληθούν κυρώσεις σε μια κυβέρνηση εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά βραχυπρόθεσμα δεν μπορούν να, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, μπορούν να τρέψουν την κατάσταση. Χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, αυτά τα οποία έχουμε, ακούσαμε και από τον Μάριο Μόντι για τη μακρυπρόθεσμη προοπτική, αλλά εν πάση περιπτώσει οι καθημερινές δραστηριότητες δεν μπορούν να υπολογιστούν με αυτόν τον τρόπο. Βράχει πρόθεσμα. Εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι είναι τουλάχιστον βράχη πρόθεσμα εξωγενείς αυτοί οι παράγοντες ως εργαλεία χάραξης πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. καθηγητή Χόρν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση του κυρίου Γκοζές. Οι αγορές ε, είναι ακόρεστες. Ζητούν όλο και περισσότερα. Μερικές φορές, ναι, και κατά τρόπο ιστερικό. Εάν δηλαδή ε, διαισθανθούν αβεβαιότητα αν κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς που είναι η κατάσταση. Αν κάποιοι θεσμοί μάλιστα τεθούν εν κινδυνό, αντιδρούν ιστερικά και, και κατά τρόπο πανικόβλητο οι αγορές και προσπαθούν να τραβήξουν τα λεφτά τους. Και αντίστροφα σε πολύ θετικέ εξελίξει βλέπουμε ότι υπάρχει υπερκάλυψη. Το είδαμε αυτό και στι ΗΠΑ και σε άλλε χώρε. Άρα, απαραίτητο είναι οι αγορέ να έχουν κάποιο πύχη αξιόπιστο ένα ορόσημο με βάση το οποίο να πούνε εάν προχωρήσουμε προς τα εκεί φτάνουμε σε κάποιο όριο, εάν προχωρήσουμε προς τα λού φτάνουμε σε κάποιο άλλο όριο. Αυτό είναι αντίστοιχα το θέμα της δομής της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Αυτό χρειάζεται δηλαδή την κρίση, την αντιμετωπίσουμε επειδή δεν υπάρχουν τέτοια ορόσημα γιατί οι αγορές διαισθάνονται ότι δεν είναι η κατάσταση ε, βιώσιμη. Δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος, δεν είναι βιώσιμο το πορτογαλικό, το ιρλανδικό και βέβαια δεν ξέρουν και τι ακολουθεί. Όσο λοιπόν δεν είναι αξιόπιστη η δομή της διακυβέρνησης, θα έχουμε τέτοιες ε, ψυχόρμητες αντιδράσεις. Και άρα χρειάζεται να θεσπιστεί το χειρότερο δυνατό μια αξιόπιστη δομή. Και αν είναι αξιόπιστη, θα σταματήσουν οι αγορές να αντιδρούν μέσα σε όρια βέβαια. Και όπως είπε και ο Πολ Τεγκράου, οι προοπτικές για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, η ιδέα των, ε, της αναδιάρθρωσης δεν θα ήταν βιώσιμες ούτε για τη Γερμανία. Βιώσιμες θα ήταν μόνο αν είχαμε ένα αξιόπιστο σύστημα. Για τον κύριο Μπούλμαν, τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο σε μια τέτοια κατάσταση. Η απάντηση θα σας δώσω είναι η εξή. Καλό θα ήταν οι προτάσεις τις οποίες υπέβαλε η Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο σίγουρα δεν ε, καλύπτουν τα όσα είπαμε εμείς εδώ ως ιδέες ε, δεν είναι δηλαδή πλήρη. και γι' αυτό θα ήταν καλό να συμπληρωθούν ώστε να αξισορροπηθούν ε, οι ε, οικονομικές ανισότητες, τα προβλήματα στις διαδικασίες, όλα αυτά τα οποία οδηγούν στα προβλήματα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση, όπως ελπίζουμε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και σε θέση να προετοιμαστούμε και να ε, οχυρωθούμε έναντι μιας προσεχούς ενδεχόμενης κρίσης. Και εδώ δεν λησμονώ φυσικά ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και όχι ένα εθνικό το οποίο προάγει τα μεν ή τα δε εθνικά συμφέροντα. Σε το πιστεύω ότι έχει σαφέστατο ρόλο να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την ανάπτυξη μιας οικονομικής διακυβέρνησης πάνω απ' όλα με ευρωπαϊκή προοπτική. Το έχει τεράστια σημασία. Δεν θα είναι μια εθνική προοπτική στηριζόμενη σε βραχυπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα, αλλά μια ευρωπαϊκή προοπτική και αυτό είναι ο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Φίλη Σιλβί Ντιέγκο. Με συγχωρείτε, ε, αλλά ε, έπρεπε να εξηγήσω την κατάσταση του Βελγίου και γι' αυτό βγήκα από την αίθουσα. Έχω δύο ερωτήσεις στον ε, καθηγητή Μανάς. Δηλαδή μπορείτε να μας εξηγήσετε το σύστημά σας βαθμολόγησης με σημεία ε, καλύτερα για τον καθηγητή Χόρν όταν ε, μιλάτε ε, για την ανάγκη ενός Ινστιτούτου που θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει ε, το, το χρέος στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι το νέο, ο νέος οργανισμός καλύπτει ε, την εποπτική δομή γιατί πιστεύω ότι αυτές οι φούσκες δημιουργούνται από τα χρέη και θα ήθελα να υπάρχει καλύτερη κατανομή εργασίας. Επίσης και προς τους τρεις σχετικά με την ε, φορολογική πολιτική και τη συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή Μόντι. Πιστεύετε ότι το ταμπού αυτό πρέπει να αρθεί και ότι χρειαζόμαστε κάποιο είδος συντονισμού φορολογικού στην Ευρώπη ή τουλάχιστον στα πλαίσια της Ευρωζώνης για να λειτουργήσει το σύστημα ή είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Σας ευχαριστώ και τους τρεις μία ερώτηση πολύ συγκεκριμένη στον κύριο Ντεγκρόστ για την οποία θα επιμείνω και ρωτώ. Στο σύστημα Red Bond, Blue Bond πώς υπολογίζουμε το επιτόκιο. Ποια είναι η αρχή που το αποφασίζει, γίνεται εκ των προτέρων, ε, γίνεται ανεξάρτητα ή είναι κάτι το πιο πολιτικό. Θέλω περισσότερες πληροφορίες. Και μετά Καθηγητή, καθηγητή Τάμενας, κάτι με ενοχλεί στο σκεπτικό σας. Εσείς ξεκινάτε με την ιδέα ότι βρισκόμενοι μέσα στην ΟΝΕ είμαστε ακόμα απόλυτα κυρίορχοι. Οπότε θα έπρεπε να αποφασίσουμε, να παρλάβουμε αποφάσεις οι οποίες πάνε, κατα, στρέφονται κατά της εθνικής κυριαρχίας Μα εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Είναι ακριβώς το αντίστροφο που αληθεύει. Βρισκόμαστε σε ένα σύστημα καταμερισμένης κυριαρχίας. Εμείς στη Γαλλία βρισκόμασταν σε μία, de facto σε μία, στη ζώνη ε, Μάρκου και κερδίσαμε σε κυριαρχία τώρα γιατί στο παρελθόν ας μου η Bundesbank αν θα έπρεπε εμείς να υποτιμήσουμε το φράγκο ή όχι. Λοιπόν, αν εμείς λοιπόν είμαστε κυρίαρχοι και θέλουμε να μας αφαιρέσουν την κυριαρχία, τότε όντως αυτό είναι δύσκολο. Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σε ένα πλαίσιο καταμερισμένης κυριαρχίας. Οπότε προς τα πού τίνει αυτός ο καταμερισμός. Ε, καταμερισμός και των φορολογικών μας. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε μέσα σε, σε μία ε, θυμική ε, απάτη όπου πιστεύουμε δηλαδή ότι όλα παίζονται στα θέματα της κυριαρχίας. Ο Διέγκο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σάρων. Εγώ είχα υποσχεθεί ότι θα είμαι σύντομο και θα κρατήσω το λόγο μου. Μία ερώτηση για όλους τους ομιλητές, τους οποίους και ευχαριστώ ειλικρινά για την τοποθέτησή τους. Η ερώτηση αφορά στο ζήτημα του χρέους. Θα ήθελα να ξέρω Τι πιστεύετε για τον κανόνα μείωσης σε δεκατημόρια αυτού του χρέους. Ο καθηγητής Μενάς ανέφερε το θέμα, συμφωνείτε με τη λογική του δωδεκατημορίου που ανέφερε ο καθηγητής. Η δε πρόταση είναι να μην γίνει σε ένα χρόνο αυτή η μείωση, αλλά σε τρία χρόνια. Και αν θέλουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, να βρούμε μια άλλη λύση. Ποια θα ήταν όμως αυτή η άλλη λύση? Ευχαριστώ. Ε, θα ακολουθήσουμε την ίδια σειρά και θα έλεγα ο Wayne ε, πέντε λεπτά περίπου, οπότε... Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Λάμπερτ σχετικά με τη φορολογία. Εάν χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό φορολογικό και ναι και όχι. Ε, αν μιλάμε για φορολογικό συντονισμό στην Ευρωζώνη μακροπρόθεσμα μπορούμε να επιβιώσουμε μόνο εάν υπάρχει μία δημοσιονομική ένωση δηλαδή να αποποιηθούμε κάποιο ποσοστό της ε, φορολογικής κυριαρχίας προς κάποια ανώτερη αρχή ε, και λέγεται ότι αυτό πρέπει να γίνει σε 20-30 χρόνια αλλά είναι απαραίτητο για να επιβιώσουμε και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ δύσκολο αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε με μικρά βήματα και να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από όλα τα προγράμματα τα οποία είναι συζήτηση τώρα. Ε, όπως είπε και κάποιος προηγούμενος ομιλητής ο οποίος είπε ότι όλα τα προγράμματα που έχουμε τώρα προς συζήτηση τόσο στερούνται φιλοδοξίας ώστε μπορούμε να προβλέψουμε ότι ε, δεν θα προχωρήσουμε πολύ για να αποφύγουμε μία επόμενη κρίση και ε, την κατάρρευση της Ευρωζώνης. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αμφιβολίες στα πλαίσια αυτά. Θα απαντήσω γαλλικά. Μα για το θέμα του υπολογισμού των επιτοκίων, με πολλούς τρόπους μπορούμε να τα υπολογίσουμε τα επιτόκια. Εγώ είχα κατά νου όμως ότι σίγουρα το επιτόκιο που εφαρμόζεται στο ευρωμόλογο θα είναι ενιαίο. Οπότε θα, υπάρχει και ένας μηχανισμός ανακατανομής στο, τμήμα, στο, στο μπλε τμήμα και θα συνδέεται με τα επιτόκια που διαπιστώνουμε στις εθνικές αγορές. Στο βαθμό δηλαδή που συνεχίζουν να υφίστανται οι εθνικές αγορές αν δεν εξαφανιστούν στο μεταξύ. Οπότε το επιτόκιο αγοράς ε, των εθνικών αγορών θα αποτελεί το δίκτυ. Πρέπει όμως να μειώσουμε το κόστος. 12% πληρώνει η Ελλάδα, 9% η Ιρλανδία. Αυτό είναι ασύλληπτο. Ας πούμε στο μπλε τμήμα τι θα γινόταν, η Ελλάδα θα συνέχιζε να πληρώνει 12% και η Ιρλανδία 9% πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό που θα αμβλύνει αυτή τη διαφορά και θα ε, καταλήγει σε μία κάποια ανακατανομή. που θα μας επέτρεπε να απαλείψουμε το πρόβλημα των χωρών 3α που φοβούνται δηλαδή ότι θα έχουν πολλά να πληρώσουν. Αυτή είναι η, βασική, η βάση που με ενέπνευσε για τη λύση του προβλήματος. Α, και του κύριου Φαγιώ. Δηλαδή να μειώσουμε το, το χρέος κατά ένα εικοστό το χρόνο ή να έχουμε μια πιο ευέλικτη ε, μέθοδο. Είμαι υπέρ μιας ε, ευέλικτης μέθοδος. Αντιλαμβάνουμε ότι, και ο καθηγητής Μανάς σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, πρέπει όμως να είμαστε ευέλικτοι. Και ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να τονίσω τώρα, άπαξ και έχω το λόγο, είναι ότι υπάρχει υπάρχει μία έμονη ιδέα στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή σχετικά με τα δημοσιονομικά προβλήματα. Όπως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ήταν καταρχήν ένα πρόβλημα υπερβολικών χρεών και ελλημάτων. Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι ισχύει με την, και ότι έχει κάποια σχέση με την κρίση ε, η, κρίση αυτή οφείλεται με μία συσσόρευση ιδιωτικού χρέους στο παρελθόν εκτός από την Ελλάδα και όχι δημοσίου. Άρα δεν χρειαζόμαστε τη σταθερότητα την οποία πρεσβεύεστε γιατί ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ δεν έχει σχέση με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και γι' αυτό θεωρώ ότι η επιβάλλουμε η υπερβολική ε, ε, ε, αυστηρότητα που δεν λύνουν τα δημοσιονομικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με τις τελευταίες παρατηρήσεις για την αρχή της κρίσεως για τα διάφορα κράτη. Ε, υπάρχουν κράτη όπου υπάρχει, υπήρχε ένα πλεόνασμα και μετά υπήρξε μία συσσόρευση χρεών λόγω της υφέσεως. Απ' την άλλη πλευρά όμως όντως ισχύει ότι στις ευρωπαϊκές χώρες το χρέος είχε αρχίσει να αυξάνεται έστω και λίγο πριν την κρίση και στο, στο σύστημα αυτό το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης δεν λειτουργεί και εφόσον υπάρχουν ποσοστά πάνω από 8% πρέπει να δούμε πώς θα επανέλθουμε σε μια σταθερή κατάσταση. Ας προχωρήσω όμως πέραν αυτών των σχολείων στο πρώτο ερώτημα του κυρίου Λομπέρ σχετικά με το σύστημα βαθμολόγησης με σημεία και έχω ένα σύντομο έγγραφο που είχε δημοσιευθεί εις το δελτίο του προσωπικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2007 και όπου παρουσιάζεται η εξής ιδέα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, εξασφαλίσουμε να υπάρχει μία δημοσιονομική πειθαρχία, δηλαδή ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός και συγχρόνως για να το επιτύχουμε ε, δεν πρέπει να αποποιηθούμε την σταθερότητα. Πώς λοιπόν θα υπάρχει πιο ευέλικτο σύστημα. Θα πρέπει σε περίπτωση που υπάρχει υψηλό χρέος μίας χώρας θα δούμε ποια είναι τα πλεονάσματα προπολογισμού που χρειάζεται για να είναι βιώσιμο το σύστημα και μετά προβαίνεται στις αναγκαίες ε, τροποποιήσεις και προσαρμογές και αν η χώρα κάνει κάτι παραπάνω, δηλαδή ε, αν κάνει 2% παραπάνω από ό,τι έκανε τότε έχει ένα πιστοτικό υπόλοιπο για να κάνει κάτι λιγότερο σε δύσκολη περίοδο. Και κατά μέσον όρων, κατά αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να θεωρήσετε ότι η πολιτική σας είναι βιώσιμη, αλλά το κράτος έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περισσότερο σε κακές εποχές και να προσαρμοστεί περισσότερο σε καλές εποχές που είναι ακριβώς αυτό που επιζητείτε. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι θέλετε ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο θα εξασφαλίσει ότι γενικώ ε, θα καταλήξετε σε μία βιώσιμη πολιτική. Αυτή είναι η ιδέα μου. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της κυρίας Γκουλάρ, ίσως δεν διαφωνώ μαζί σας σχετικά με την κυριαρχία και αν πρέπει να υπάρχει μια κατανομή μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης αλλά οι παρατηρήσεις μου αναφέρονται πιο πολύ στο τι θα, πού πρέπει να τεθεί ο πύχης όπως είπατε και προηγουμένως ο Μέλαμπαρ και ε, πιστεύω ότι ο πύχης αυτός θα έπρεπε ε, να βρίσκεται στο επίπεδο του συντονισμού και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Φεγιό με συγχωρείτε αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας σχετικά με τον κανόνα μειώσεως 8% που πρότεινε ε, το περασμένο Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κριτική μου στην πρόταση αυτή ουσιαστικά αναφέρεται σε τρία σημεία, διότι ε, οι περισσότερες χώρες εκτός ελαχίστων τώρα βρίσκονται πάνω από το 60% και οι περισσότερες ε, υπερβαίνουν και το 80% του ΑΕΠ, τότε η εφαρμογή ενός τέτοιου κανόνα θα ε, απαιτούσε μία συντονισμένη συρρήκνωση όλων των κρατών της Ευρώπης. Οπότε τότε ο, συντελεστή ο συντελεστής πολλαπλασιασμού είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αν πρόκειται για ένα κράτος και η ε, επίδραση αυτής, αυτού του του κανόνα στην ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Δεύτερον, έχουμε ήδη ένα νόμισμα για όλους ε, το οποίο να αμφισβητείται από πολλούς αλλά αυτό που δεν θέλετε είναι να ισχύσει ο ίδιος κανόνας για όλους διότι έχουμε ανισορροπίες μεταξύ κρατών και αν έχετε μια χώρα σαν την Ισπανία ή την Ιρλανδία που έχει μεγάλο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών και μετά τη Γερμανία που έχει μεγάλο πλεόνασμα, τότε ε, αν ε, αυτές οι χώρες συρρυκνωθούν η κατάσταση θα είναι πιο δυσχερή σε άλλες χώρες. Θέλετε λοιπόν κάποια ευελιξία ώστε οι χώρες με πλεόνασμα να συνεχίσουν επεκτατικές πολιτικές και οι χώρες με, ε, με συρρήκνωση να έχουν περιοριστικές πολιτικές. Αλλά να μην υπάρχει το ίδιο σύστημα για όλους διότι στις χώρες που υπάρχει μεγάλο χρέος ε, ε, χρειάζεται μία πολύ αυστηρή ε, φορολογική πολιτική. Πρέπει να γίνουν ορισμένοι υπολογισμοί και θα δείτε βάσει του εγγράφου που σας έχω μοιράσει ότι για τα επόμενα 20-30 χρόνια εάν έχουμε κάποιο επίπεδο επιτοκίων στην Ιταλία θα πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα επιτόκιο 5% το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό. Λοιπόν, ε, η έλλειψη της αξιοπιστίας είναι σημαντική διότι ε, αυτοί οι κανόνες δεν μπορούν να ισχύσουν. Ευχαριστώ. Ναι, ρωτήσατε για την κατανομή εργασίας ως προς την αντιμετώπιση του υπερβολικού πλεονάσματος. Μάλλον των υπερβολικών ανισοζήτων ανισοτήτων. Ναι, υπάρχουν λύσεις, όπως η παραδείγματι κατανομή εργασίας προς το εξή ότι το ένα όργανο επιτηρεί, εποπτεύει, εντοπίζει προβλήματα, το άλλο πυροσβεστικά έρχεται για να κατασβέσει τα προβλήματα την ώρα της κρίσης. Αυτό είναι μια λύση ως προς το θέμα της κατανομής εργασίας. Επίσης, για να περάσω στη τελευταία ερώτηση πριν ξαναγυρίσω κάποιες άλλες, μια πρόταση της Επιτροπής για μείωση του χρέους. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για οικονομικό πρόβλημα. Δεν είναι μηχανικό το πρόβλημα. Δεν είναι μηχανολογικό μάλλον. Άρα πρέπει να είναι κανείς ευέλικτος. Ιδάλλως, εάν το λύσουμε μηχανιστικά, αυτό που ανέφερε και ο καθηγητής Μανάς ουσιαστικά, θα έχουμε υπερβολική δημοσιονομική συρρήκνωση στην Ευρωζώνη και όπως είδαμε και στην κρίση το 2009, όπου όλες οι χώρες θέσπισαν πακέτα κινήτρων, οι δικοί μας υπολογισμοί με θετικούς τότε δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές συνόδευαν αυτήν την κρίση σε σχέση με, ένα, με μια υπόθεση όπου οι χώρες θα ακολουθούσαν η μία την άλλη, θα προχωρούσαν ε, διαδοχικά δηλαδή στην ε, φάση αυτή. Αν όμως πάνε ταυτόχρονα όλες οι χώρες, οι ε, συνέπειες είναι βέβαια πολλαπλάσιες. Εδώ λοιπόν μια προσέγγιση ευέλικτη από το Συμβούλιο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, ε, Ιρλανδία μάλλον, ε, Πορτογαλία που έχουν σημαντικά ε, ελλείμματα, θα πρέπει μάλλον να περάσουν σε πιο, από πιο στενά μονοπάτια. Ενώ οι άλλες χώρες που δεν έχουν ακόμη το σοβαρό πρόβλημα θα πρέπει να περιορίσουν τις δαπάνες τους ώστε να ικανοποιήσουν την ανάγκη για δημοσιονομική λιτότητα που γεννούν οι άλλες χώρες. Γιατί τα δημοσιονομικά της ζώνης του ευρώ δεν είναι και τόσο λαμπρά γενικά. Να τα συγκρίνουμε με τις ΗΠΑ για παραδείγμα, όπου από όπου ακούγονται πολλές, για την ισχύουσα κατάσταση. Για τη Γερμανία χωρί τη Γερμανία μάλλον, οι προβλέψει μα για, την, για ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ είναι 0,6% χωρί τη Γερμανία. Πολύ χαμηλή. Άρα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να προχωρήσει σε ανάκαμψη εγκαίρω όπω θα θέλαμε και με βάση προβλέψει που είχαν προηγήθει τη κρίσεω. Και άρα δεν μπορούμε να ανθέξουμε οικονομικά αυτή την κρίση χωρί μια σημαντική δημοσιονομική αναδιάρθρωση. Αυτό όμω θα πρέπει να το κάνουν οι χώρε εκείνε που έχουν πλεόνασμα. Όχι αυτέ οι οποίες έχουν έλλειμμα δεν μπορούν να το πράξουν οι χώρες που έχουν έλλειμμα, δεν αντέχουν να το πράξουν. Και άρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να υποστεί τα ίδια μέτρα η κάθε χώρα, δεν θα περάσει κάθε χώρα από τη δημοσιονομική αναδιάρθρωση, άλλες είναι υποχρεωμένες να το κάνουν, άλλες δεν θα πρέπει να ε, υποχρεωθούν να το πράξουν. Και έχουμε τώρα μια πολύ ουσιαστική ερώτηση ως προς την ανεξαρτησία στην Νομισματική Ένωση πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Ή θα συρθούμε σε μια απόφαση διαφορετικά. Η απόφαση είναι τι θέση έχουμε, τι είδους ανεξαρτησία έχουμε τώρα, είτε θεωρητική είτε πρακτική, και τι είδους κανόνες και ρυθμίσεις μπορούμε να επιβάλλουμε στις διάφορες κυρίαρχες χώρες, προκειμένου να τους υποχρεώσουμε να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή να μην, έχουν τον, ε, να μην έχουμε μέσο πληθωρισμό άνω του 2%. Δηλαδή ώστε να μην ξαναπέσουμε σε κατάσταση σημαντικής ε, ε ανισορροπίας των ισοζυγίων των συναλλαγών. Ή πώς μπορούμε ενδεχομένως να προχωρήσουμε προς μια περισσότερη οικονομική ένωση, ολοκλήρωση δηλαδή, με ε, εγκατάλειψη, με εκχώρηση αρμοδιοτήτων με εκχώρηση κυριαρχία ουσιαστικά προς κάποια όργανα θεσμικά, τα οποία θα μπορούν σχετικά αυτόματα να ε, ρυθμίζουν, να διορθώνουν τις ανισορροπίες. Αυτό το δεύτερο θα προτιμούσα εγώ βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό πολιτικά στα επόμενα χρόνια. Πάντως, εν ευθέτω χρόνο, θα ανακαλύψουμε ότι απαιτείται ο ελάχιστος τουλάχιστον συντονισμός, ώστε να έχουμε να μην έχουμε καλύτερα dumping είτε φορολογικό είτε κοινωνικό είτε μισθολογικό. Αυτός ο ελάχιστος συντονισμός απαιτείται. Ιδάλλως, τελικά, κινδυνεύουμε να παραβούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ε, σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης. Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος και ε, τους ομιλητές ιδιαίτερος και βέβαια τον καθηγητή Μόντι που έκανε την κύρια εισήγηση νωρίτερα. Ευχαριστώ τους βουλευτές ε, που έδειξαν την αντοχή και έφτασαν μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως. Οι παρουσιάσεις έχουν διανεμηθεί στους συναδέλφους και πάλι μπορούν να σας αποσταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν το προτιμάτε, ώστε να τις διατηρήσετε στο αρχείο σας. Δεν μου μένει παρά να σας ευχαριστήσω και πάλι και να κηρύξω το πέρα της συνεδριάσεως λίγο νωρίς.